Liebe Kolleginnen und Kollegen, Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω να ξεκινήσουμε. Δεν έχει γεμίσει βέβαια ακόμα η αίθουσα, αλλά νομίζω ότι ε, κατά τη διάρκεια του πρωινού θα αλλάξει αυτό. Σας καλωσορίζω λοιπόν στην ε, σημερινή συνεδρίαση και χαίρομαι πραγματικά που μπορώ να σας καλωσορίσω στην ε, Ολομέλεια της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής μας για το θέμα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο θέμα αυτό αφιερώθηκαν ήδη χτε ε, τρει παράλληλε συνεδριάσει ε, με πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα. Αυτά τα πάνελ ε, θα τα ξαναδούμε βέβαια σήμερα, όχι μόνο θεματικά, αλλά και οι πρόεδροι των τριών πάνελ, η συνάδελφοι Σίλβια Κώστα, ο κύριος Διάκονου και η Σαμπίνε Φερχάγεν, ε, θα μας κάνουν μια σύντομη παρουσίαση για τις συζητήσεις που διεμήθησαν στα τρία πάνελ, έτσι ώστε να έχουμε όλη μια ιδέα γενική για το τι συζητήθηκε στις άλλες ομάδες που δεν ήμασταν παρόντες. Επίσης είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σήμερα διαφορετικά από χτες, όπου ε, μπορέσαμε να το έχουμε αυτό μόνο για μία, ε, σε μία συνεδρίαση, έχουμε, έχουμε διερμηνία και σε όλες τις επίσημες γλώσσες και χαίρομαι πραγματικά που η σημερινή ε, ε, διάσκεψη ε, γίνεται υπό την αγίδα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντώνιο Ταγιάννη, και αυτό υπογραμμίζει πραγματικά την μεγάλη σημασία που δίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Έτο πολιτιστική Κληρονομιάς, αλλά και στην ανταλλαγή ιδεών με τα Εθνικά Κοινοβούλια Παρόλο που ο πρόεδρο Ταγιάννη δυστυχώ δεν θα μπορέσει να είναι παρόν σήμερα έχει κάποιε άλλε ανηλυμένε υποχρεώσει και πρόσφατα κύρωσε την ε, συμμετοχή του. Ε, τις τελευταίες ημέρες γιορτάσαμε τα 100 χρόνια από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και πραγματικά αυτό μας θυμίζει και την, ε, ε, τον πολυσχηδή χαρακτήρα του ευρωπαϊκού, της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και τις προκλήσεις που αυτή μας δημιουργεί. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω κάποια σχόλια για το θέμα αυτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις, ίσως τις μεγαλύτερες από ποτέ, από την ιστορία της. Οι οικονομικές ανασφάλειες, κυρίως ε, λόγω των ε, διεθνών εμπορικών σχέσεων που συνεχώς αλλάζουν, ένα ε, διεθνές πεδίο που πλήττεται από συγκρούσεις, από δυσλειτουργία και από αλλαγή στι παγκόσμιες ε, σχέσεις δυνάμεων, επίση, οι μεταναστευτικέ ροές ε, και τα προβλήματα που απορρέουν σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση, αλλά και οι σημαντικές συζητήσεις που γίνεται για το σήμερα αλλά και για το αύριο της ευρωπαϊκής, ε, του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, διέπουν την ε, σημερινή συζήτηση στην Ευρώπη και την πραγματικότητά τη. Βλέποντα λοιπόν αυτέ τις ε, προκλήσεις, πολλοί μπορεί να τίνουν να θεωρούν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολιτική προτεραιότητα, ούτε βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ το εξή. Ο πολιτισμό είναι το πιο σκόπιμο και το πιο αποτελεσματικό ε, ε, μέσο για να μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσει ε, στα ερωτήματα για το μέλλον της Ευρώπη και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση στην Ήπειρο που ε, όντως δημιουργεί μια βαθιά κρίση ταυτότητα. Για να δείξουμε ποια είναι αυτή η κρίση πρέπει να θέσουμε τρία ερωτήματα. Ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε. Αυτά τα τρία βασικά θεμελιώδη ερωτήματα ήταν και τα βασικά κίνητρα ε, τα οποία διήψαν το, το Ευρωπαϊκό Έτος της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 παρά τις αρχικές ε, δυσκολίες που αντιμετώπισε τελικά στο τέλος του με συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στηρίχθηκε από πολλές ε, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και μπόρεσε να τελεσφορήσει. Και το Ευρωπαϊκό Κέντρο της, το Ευρωπαϊκό ε, έτος της ε, πολιτιστικής κληρονομιάς δεν είναι ευρωπαϊκό μόνο γιατί το λέει το όνομά του, αλλά ακριβώς επειδή είναι φιλόδοξος προς αυτό. Το έτος που τελειώνει σιγά σιγά θέλει να, προσπεράσει τα εθνικά και τα γλωσσικά σύνορα και να θεωρήσει τον πολιτισμό ως ένα δεσμό του ευρωπαϊκού πολιτισμού για να μπορέσουμε να συνδέσουμε όλες τις επιτυχίες του... της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό ισχύει και ως προς τη χρονική στιγμή και γι' αυτό ε, το, μότο αυτής της, αυτού του έτους είναι πραγματικά πάρα πολύ σωστό. Η κληρονομιά μας εκεί που το παρελθόν συναντά το μέλλον. Η σημερινή διάσκεψη θα μας βοηθήσει ε, από κοινού ως πολιτικοί και ως πολίτες να συζητήσουμε και να αναλογιστούμε τις διάφορες ε, πτυχές και το δυναμικό της πολιτιστικής κληρονομιάς. Γιατί η πολιτιστική μας κληρονομιά θα πρέπει και μετά το 2018 να αποτελέσει μια κεντρική αξία στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής και μάλιστα κυρίως επειδή αποδείχθηκε ότι είναι παραπλανητικό να θεωρούμε ότι μόνο ένα ευρωπαϊκό οικοδόμημα που βασίζεται σε οικονομικές στεναρές βάσεις μπορεί να αντιμετωπίσει όλες τις ε, κρίσεις που προκύπτουν και να εγγυηθεί το ότι οι πολίτες μακροπρόθεσμα θα ταυτιστούν με τον όρο Ευρώπη. Όπως έχουμε, έχει υποθεί πολλές φορές, και όπως έγινε και, το, τον προηγούμενο Δεκέμβρη στο Μιλάνο όταν ξεκίνησε το έτος πολιτικής κληρονομιάς αλλά και τον Ιούνιο με την διάσκεψη που κάναμε με τον πρόεδρο Ταγιάννη και τον πρόεδρο Ιού, ε, Γιούνκερ με τίτλο «Πολιτιστική κληρονομιά στην Ευρώπη». Ε, δεν θέλω να δημιουργήσω μια αφελή αισιοδοξία σήμερα. Μια αισιοδοξία η οποία θεωρεί ότι το, ο πολιτισμός είναι η πανάκια για όλα τα προβλήματα της Ευρώπης ή για όλα τα προβλήματα του κόσμου όπως κάθε τι ανθρώπινο και ο πολιτισμός ε, έχει ε, εγγενή στοιχεία αμφισημίας. Μπορεί να δημιουργήσει, να απελευθερώσει αρνητικές και θετικές ενέργειες, μπορεί να είναι συγκολητική δύναμη αλλά και διασπαστική, μπορεί να ε, καταρρύψει σύνορα, μπορεί και να υψώσει σύνορα. Και το τελευταίο συμβαίνει όταν ο πολιτισμός θεωρείται μέσω σοβινισμού, αποκλεισμού, δυσφήμισης του ενός ή του άλλου ο πολιτισμός είναι αυτός που μας διαχωρίζει, ε, μας, διαφοροποιεί, αλλά δεν είναι κάτι που μας χωρίζει, είναι κάτι που μας ενώνει. Από, χώρα, από τις χώρες ως τις πόλεις, από το ένα κράτος μέλος ως το άλλο, από το παλιό στο νέο, από το παρελθόν στο μέλλον. Και έτσι ο αγώνας για τον πολιτισμό θα πρέπει να γίνει με, θετική, με θετικό πρόσημο και να μην ε, τον αντιμετωπίσουμε ως ε, μια υποκουλτούρα, όπως ανέφερε και ο ιστορικός συγγραφέας Καλ Κράους πριν από 100 χρόνια. Είναι πολύ σημαντικός ο στόχος αυτός και η πολιτιστική κληρονομιά ζητά μια σταθερή προσπάθεια. Αυτή την ε, κληρονομιά να την κατανοήσουμε, να τη διατηρήσουμε, και να την εγγυηθούμε και για το μέλλον. Όπως λέει και ο ε, Γκέτε στον ε, Φάουστ, ότι κληρονομεί κανείς από τους ε, ε, γονείς του πρέπει να το κάνει δικό του για να μπορεί να το αποκτήσει. Χαίρομαι λοιπόν πολύ κυρίες και κύριοι που ε, θα μπορέσουμε σήμερα και αυτή την, αυτό το ανοιχτό πνεύμα να το προωθήσουμε αλλά και την προσπάθεια αυτή ώστε οι πολίτες να δούνε και το καλύτερο που μπορεί να τους προσφέρει η Ευρώπη και ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Πάμε τώρα στη, στους γύρους της συζήτησης και στις διάφορες παρεμβάσεις. Καταρχάς, έχουμε πάρα πολλούς ομιλητές σήμερα. Οπότε, ο στόχος της α, ε, σημερινής διάσκεψης είναι να μάθουμε από τις εμπειρίες των κρατών μελών ώστε να έχουμε μια ε, καρποφόρα ανταλλαγή απόψεων. Οπότε, εγώ θα κλείσω την ε, δική μου παρέμβαση και πριν δώσω το λόγο στους άλλους ομιλητές να σας αναφέρω λίγο τα χρονικά όρια γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικά για τη σημερινή συζήτηση ο χρόνος αγόρασης θα τηρηθεί ευλαβικά. Οι συνάδελφοι από την ε, Επιτροπή ε, ε, Πολιτισμού ξέρουν ότι μπορώ να είμαι πολύ αυστηρή. Αν έρχεται, φτάνει στο τέλος ο, χώρος, ο χρόνος αγόρευσής σας, θα αρχίσω να χτυπάω το σφυράκι μου. Γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι και στον επόμενο που θέλει να πάρει το λόγο. Οπότε θα προσπαθήσω όλους να σας ε, υποχρεώσω σε εισαγωγικά να τηρήσετε τον χώρο, το χρόνο αγόρευσης γιατί αλλιώς θα μιλάμε αενάως. Και κάποια στιγμή θα χάσουμε και τους διερμηνείς. Οπότε, ο χρόνο αγόρευσης, όπως είπα, θα τηρηθεί ευλαβικά και βεβαίω θα δούμε ανάλογα και με τον ε, αριθμό των ομιλητών πώς θα τα οργανώσουμε, πώς θα τον κατανείμουμε. Το πολύ δύο λεπτά όμως θα δώσω στον καθέναν. Οπότε να το έχετε υπόψη σα. Μετά, οι ε, βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων που θέλουν να πάρουν το λόγο παρακαλούνται να συμπληρώσουν το έγγραφο που υπάρχει μπροστά σας. Πρέπει να ε, το έχετε όλοι και να μας πείτε σε ποιο πάνελ θέλετε να πάρετε το λόγο. Και στο τέλος του κάθε πάνελ και με την, μετά την ε, περίληψη από τα τρία θεματικά πάνελ θα γίνει μια συζήτηση με ερωταπαντήσεις και βεβαίως θα δούμε πόσο χρόνο θα έχουμε γι' αυτό ανάλογα και με τις ε, ερωτήσεις και τους ε, ομιλητές που θέλουν να πάρουν το λόγο. Τώρα, ε, με μεγάλη μου χαρά θα δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της Αυστριακής Προεδρίας, την ε, ε, πρέσβη κυρία Elizabeth Κόνφαϊντ. Μετά θα ακούσουμε την κυρία Θέμιδα Χριστοφίδου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας κάνει μια παρουσίαση. Καταρχάς θα ακούσουμε όμως την κυρία Κόνφαϊντ και καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, αγαπητοί βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας μιλήσω για τους βασικούς στόχους της Αυστριακής Προεδρίας στα πλαίσια του πολιτιστικού έτους. Ε, αυτό το έτος πολιτιστικής κληρονομιάς, το 2018, είναι, ένα από τους, είναι ένας από τους βασικούς στόχους της ε, Αυστριακής Προεδρίας. Ταυτόχρονα ξέρουμε πόσο μεγάλη σημασία δίνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε, την αφορά, και σε ό,τι αφορά την ε, εξαγωγή συμπερασμάτων, αλλά και στην εφαρμογή σημαντικών πρωτοβουλειών. Η μεγάλη δέσμευση από πλευρά του Κοινοβουλίου πραγματικά εκτιμάται ιδιαίτερω από το Συμβούλιο η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κληρονομιά δεν, δεν υπάρχει από μόνη τη. Είναι ένα πολύ σημαντικό οικονομικό, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό πόρο, ο οποίο ε, μπαίνει τώρα στο προσκήνιο. Μπορεί να βοηθήσει στην ε, καλύτερη δόμηση του ε, μέλλοντος, μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών, μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική συνεργασία και την ε, συνοχή του κοινωνικού ιστού. Υπάρχουν πολλά project και εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη που ακριβώς ε, δείχνουν την ε, λειτουργία αυτή του πολιτισμού και μας δείχνουν την αξία του. Δημιουργείται λοιπόν μια ενσυνείδηση για τον πολιτισμό και ιδιαίτερο σημαντικό, πέραν των παραδοσιακών ιδεών που έχουμε, βλέπουμε τον πολιτισμό και ε, στο σήμερα αλλά και με όραμα στο μέλλον. Και γι' αυτό θα πρέπει να φτάσουμε σε όλους τους πολίτες, κυρίως όμως τους νέους. Εκεί προσπαθούμε να δημιουργήσουμε καλύτερη συνειδητοποίηση και να τους συμπεριλάβουμε περισσότερο. Υπάρχει ένα πόρταλ από την Αυστριακή Προεδρία που δείχνει τα τελευταία στοιχεία ε, για τις διάφορες ε, δραστηριότητες που έχουν ήδη γίνει και που προβλέπεται να γίνουν και αποτελεί βεβαίως πλατφόρμα για διάφορα project, τα οποία μπορούν να ε, διεξαχθούν, αλλά και για πρωτοβουλίες που μπορούν να προταθούν. Περίπου 186 project βρίσκονται αυτή τη στιγμή εν εξελίξη. Στα πλαίσια της, Ευρωπαϊ... της Αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου, βεβαίως, θα δείτε και κάποιες θεματικές διασκέψεις. Ε, ένα παράδειγμα θα ήθελα να σας αναφέρω εδώ. Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για την πολιτική, για την αρχιτεκτονική ε, δόμηση υψηλής ποιότητας για την Ευρώπη για όλους. Από τις 13 ε, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου διεξήχθη. Στη διάσκεψη αυτή συζητήθηκε το θέμα πώς η δόμηση υψηλής ποιότητας μπορεί να, να είναι καθημερινότητα για όλους και πώς μπορούν σε εθνικό επίπεδο να γίνουν διάφορα βήματα και να αναλυφθούν μέτρα ώστε αυτό να γίνει πραγματικότητα. Θα ήθελα επίσης να μιλήσω και για μία ε, διάσκεψη στη Βιέννη, την καταληκτική διάσκεψη της, ε, του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, Ευρώπη ε, για τον πολιτισμό, 6 και 7 Δεκεμβρίου. Η διάσκεψη αυτή θα ε, χωριστεί σε δύο μέρη. Στις 6 Δεκεμβρίου θα γίνει μια διάσκεψη προσβάσιμη σε όλους, η οποία θα θέσει την προσοχή σε όλα τα ευρωπαϊκά project. Αυτό θα γίνει στο κέντρο της ε, Βιέννης, οπότε περιμένουμε περίπου 500 με 600 καλεσμένους. Τη δεύτερη ημέρα θα γίνουν συζητήσεις, ομιλίες, πάνελ, ε, εργαστήρια, ομάδας εργασίας στα πλαίσια αυτής ε, της διάσκεψης. Και επίσης θα γίνει απονομή του βραβείου διδημοποίησης ε, για, διάφορες, ε, για διάφορα σχολικά project. Και βεβαίως χαιρόμαστε που με τον Υπουργό Μπλούμελ και με τον Επίτροπο Ναύρασιτς θα είστε κι εσείς πρόεδρε παρούσα. Επίσης, ο Επίτροπος Ναύρατσιτς θα παρουσιάσει το νέο σχέδιο δράσης για την πολιτιστική κληρονομιά και εδώ μιλούμε κυρίως για το θέμα της βιωσιμότητας του έτους πολιτιστικής κληρονομιάς. Για παράδειγμα, βιώσιμος τουρισμός, συμμετοχική καθοδήγηση για την πολιτιστική κληρονομιά και προκλήσεις για την διατήρησή της. Επίσης, θα πρέπει να δούμε και τα project των πρακτικών, αλλά και την συμμετοχή των νέων. Είναι σημαντικό για μας η στοχοθέτηση του έτους πολιτικής κληρονομιάς να ξεπεράσει τα θέματα αυτά που θα συζητηθούν εκείνες τις ημέρες. Ιδιαίτερα σημαντικό για μας είναι το follow-up για το ε, Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτικής Κληρονομιάς 2018, το οποίο θέλουμε να συνδέσουμε με διάφορα μελλοντικά project. Αυτή ακριβώς η βιωσιμότητα είναι μία από τις βασικές πέντε προτεραιότητες του σχεδίου δράσης για τον πολιτισμό για το 2019-2022. Και χαιρόμαστε που έχουμε καταφέρει να το θεωρήσουμε ως προτεραιότητα. Κατά διάρκεια της Αυστριακής ε, Προεδρίας έγιναν ε, πολλές δραστηριότητες για να τεθεί το πλαίσιο για την πολιτική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τον Ιούλιο εργαζόμαστε εντατικά και συζητούμε εντατικά για το σχέδιο ε, δράσης και τώρα στις 27 Νοεμβρίου θα ψηφιστεί το πρόγραμμα εργασίας από τους Υπουργούς. Τι καινούριο υπάρχει. Σημαντικό είναι το ότι επικεντρωνόμαστε σε επιλεγμένες προτεραιότητες με συγκεκριμένα και χρήσιμα αποτελέσματα και σε εποπτεία των αποτελεσμάτων, στην απαραίτητη ευελιξία, αλλά και στις ε, τροποποιημένες ε, ε, συνθήκες τις οποίες θα πρέπει να μπορούμε να απαντήσουμε για να ενισχύσουμε την εφαρμογή από τα κράτη-μέλη. Παράλληλα με το σχέδιο δράσης για την πολιτική κληρονομιά της Κομισιόν υπάρχουν διάφορα μέτρα τα οποία έχουν συμφωνηθεί και που προωθούν την ανταλλαγή μεταξύ των κρατών μελών και την ανάπτυξη στρατηγικών προσεγγίσεων. Μεταξύ άλλων, ενισχυμένη προσέγγιση των εμπειρογνωμόνων ε, της Ευρώπης ε, για την, ε, για την κουλτούρα και τον πολιτισμό και σε ό,τι αφορά τη δόμηση. Επίσης, εναλλακτικέ πηγές χρηματοδότησης για την πολιτιστική κληρονομιά ποιοτικά πρότυπα για την αποκατάσταση ιστορικών κτηρίων στα πλαίσια του, των διορθωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, συμμετοχική διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ό,τι αφορά την Σύμβαση Φάρο και μεταφορά τεχνογνωσίας με επισκέψεις και γενικότερη διαδικτύωση της Ευρώπη Αλλά ένα σημαντικό κομμάτι έχει να κάνει με την πρόταση της Κομισιόν Creative Europe, Δημιουργική Ευρώπη, η οποία παρουσιάστηκε στις 30 Μαΐου και από τον ε, Ιούνιο συζητείται στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Αυτό το πρόγραμμα είναι καινούριο για, την, ε, για, το, για τον πολιτισμό και την δημιουργική βιομηχανία και αποτελεί ένα σημαντικό στόχο της Προεδρίας. Ε, ο στόχος μας είναι να έχουμε σύντομα μεγάλη πρόοδο. Και στο Συμβούλιο θα υποβάλουμε μια σχετική έκθεση. Παράλληλα με αυτό ξέρουμε ότι ο φάκελο για το ε, τυχάνει διαπραγμάτευση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευχαριστώ τους ε, ευρωβουλευτές, την κυρία Κώστα για τη δέσμευση που έδειξε και σας συγχαίρουμε για την ε, επιτυχή υποβολή της έκθεσης σα τέλο Οκτωβρίου. Η πρόθεση της πολιτικής κληρονομιάς παραμένει βασικό, ε, βασικό σημείο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά project ε, που ε, χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια και μου έρχεται στο νου ήδη το 2018 ε, ο διαγωνισμός για την ενίσχυση της, συνειδητοποίηση συνειδητοποίησης και την ευρωπαϊκή κληρονομιά και τις αξίες που τρέχει μέχρι, το 2000, μέχρι το, τα μέσα του Δεκεμβρίου. Η πολιτική κληρονομιά βεβαίω δεν σημαίνει ότι ξεχνούμε την, ε, τις νέες ε, τεχνολογίες και την καινοτομία. Στις 8 και 9 Οκτωβρίου έγινε στην ε, Βιέννη μια συνάντηση εμπειρογνωμόνων με τίτλο Challenging the Content στην, το ψηφιακό περιεχόμενο στην Ευρώπη. Περίπου 360 εμπειρογνώμονες συμμετείχαν σε αυτή τη διήμερη συνδιάσκεψη με συζητήσεις για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις βασικές προκλήσεις στην ψηφιακή εποχή για την δημιουργική βιομηχανία. Ε, στο κέντρο βρέθηκε το ερώτημα πώς, μπορούμε, πώς μπορούν οι πάροχοι περιεχομένου, Ευρωπαίοι και μη, να ε, συνεργαστούν με την ε, βιομηχανία μουσικής, κινηματογράφου, πώς μπορούν να υποφεληθούν και πώς όλα αυτά μπορούν να είναι διαφανή. Η ψηφιακή οικονομία δίνει τις δυνατότητες και με τις υπηρεσίες της να δημιουργηθούν νέες, δημιουργι... νέες δυνατότητες διάχυσης περιεχομένου και αυτό σημαίνει σημαντικό δυναμικό και οικονομικό αλλά και πολιτιστικό. Ταυτόχρονα υπάρχουν σημαντικές συζητήσεις που πρέπει να γίνουν για τη διαφάνεια, για, την, για τον πλουραλισμό στα ΜΜΕ και για την πολιτιστική ποικιλία. Η διάσκεψη αυτή έδειξε ότι σε σχέση με τις βασικές αλλαγές που γίνονται στην, στο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η, τα προβλήματα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ε, συζητήθηκαν και τα εμπόδια, συζητήθηκαν και οι διάφορες στρατηγικές. Πολλά υποσχόμενες προσεγγίσεις δείχνουν την, το, το, το σύνδεσμο μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών συμπράξεων. Ε, το κοινό μάρκετινγκ και τις πλατφόρμες περιεχομένου. Οι συζητήσεις επίσης έδειξαν ότι Γενικώ ε, υπάρχει ομοφωνία ότι οι, ε, οι συνθήκες για τον ανταγωνισμό πρέπει να είναι ίσες για όλους. Αυτές οι online πλατφόρμες επίσης που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη είναι σημαντικές και θα πρέπει να τηρούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Ήδη μιλήσαμε για το θέμα της, ε, των νομικών, ε, του νομικού αντικτύπου που έχουν αυτές οι ε, πλατφόρμες και πώς μπορούμε να τις καταστήσουμε υπόλογες. Ένας, ένα έτος πολιτικής κληρονομιάς, τι θα ήταν όμως χωρίς συγκεκριμένες εμπειρίες πολιτιστικές, πώς θα μπορούσε να γίνει χωρίς να έχουμε αντίστοιχες διασκέψεις εδώ στις Βρυξέλλες. Έχουμε το πρόγραμμα πλαίσιο στις Βρυξέλλες, όπου η ε, Αυστρία παρουσιάζεται ως χώρα πολιτισμού και η Βιέννη βεβαίως και βεβαίως σας ε, καλούμε να δείτε την έκθεση αυτή και πώς μπορούν να, ε, συνεργαστούν, να συνδυαστούν οι παραδοσιακές προσεγγίσεις και η σύγχρονη τέχνη. Μπορείτε να έχετε μια διαφορετική οπτική. Και με το Μποζάρ πραγματικά βρήκαμε μια πάρα, ένα πάρα πολύ καλό εταίρο. Ελπίζω ότι μπόρεσα να σας δώσω έτσι μια γενική εικόνα για τις δραστηριότητες της Αυστριακής Προεδρίας στα πλαίσια του ε, Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Εγώ ευχαριστώ την πρέσβη. Πάμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην κυρία Χριστοφίδου. Έχετε το λόγο. Δέκα λεπτά το πολύ και εσείς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητή Πέτρα, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Εθνικών Κοινοβουλίων, συνάδελφοι. Είναι μεγάλη μου χαρά που σας μιλώ σήμερα. Γνωρίζω ότι πολλοί από εσά ταξιδέψατε από μακριά για να βρίσκεστε εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Κατά τη διάρκεια των σημερινών συζητήσεων θα συζητήσετε τρία θέματα μεγάλη σημασία και αξίας το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτικής Χρονομιάς, Πολιτική ταυτότητα, διατήρηση, συντήρηση ε, και αποκατάσταση πολιτικής χρονομιάς και την πολιτική κληρονομιά στην εκπαίδευση. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να σας πω ποιες είναι οι δικές μου σκέψεις και τι έχουμε καταφέρει να πετύχουμε μαζί αυτή τη χρονιά. Το ευρωπαϊκό έτος είναι ήδη μεγάλη επιτυχία, πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Τα νούμερα είναι εύγλωτα, πάνω από 11.000 εκδηλώσεις έλαβαν χώρα το 2018 για να γιορταστεί η πολιτιστική μας κληρονομιά. Φτάσαμε σε 6 εκατομμύρια άτομα. Ε, χωρίς την ε, στήριξη και την ε, επιμονή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα έχει γίνει πραγματικότητα αυτό το έτος και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω γι' αυτό. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω τα κράτη-μέλη που υιοθέτησαν αυτή την πρωτοβουλία μας και έφεραν ξανά στην κοινή γνώμη την συνείδηση αυτό δηλαδή που μας κάνει όλους Ευρωπαίους. Ο Επίτροπος Ναυρασίτς θα μιλήσει περισσότερο για τις επιτυχίες αυτού του έτους, αλλά αυτές οι επιτυχίες έγιναν δυνατές ε, μέσω της συμμετοχής όλων των πολιτών σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολιτικές οργανώσεις, σχολεία, μουσεία, πόλεις και περιφέρειες συμμετείχαν. Πολλοί από τους εκπρόσωπούς τους είναι εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα κάνατε. Οι δραστηριότητες του φετινού έτους έγιναν αποκεντρωμένα σε συνεργασία, στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη, καθώς επίσης και με ένα ε, ευρύ φάσμα πολιστικών οργανώσεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής των Εμπλεκομένων, των stakeholders, ε, που ανέλησαν την ε, σχέση ανάμεσα στην κοινότητα και την, στην πολιτική ταυτο, ε, ε, και την ταυτότητα. Αυτό το θέμα ήταν στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας φέτος. Πώς δηλαδή εμείς ο καθένας από εμά εκφράζει πολιστικά τον εαυτό του. Αυτή η έκφραση αποτελεί καθρέφτη της ταυτότητάς μας. Μουσική, χορή, λογοτεχνία, παραδόσεις μας ορίζουν. Το έτος αυτό δεν ήταν απλώς ευκαιρία να ξαναδούμε ποιοι είμαστε εμείς οι Ευρωπαίοι τον 21ο αιώνα, αλλά και να αναλύσουμε τις ιστορικές και πολιστικές δυνάμεις οι οποίες διαμόρφωσαν τις ε, παραδόσεις μας και την θέση μας σε αυτή την Ήπειρο. Ε, συμμετείχα σε πολλές από τις συναντήσεις, από τις εκδηλώσεις που έγιναν σε όλα τα κράτη-μέλη και είδα πολλά. Τι έγινε λοιπόν για να στηριχθεί αυτό το έτος. Διπλασιάσαμε τη χρηματοδότηση για τις ε, μέρες πολιτικής κληρονομιάς. Ε, αυτό το πρόγραμμα σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης ανοίγει τις πόρτες πολλών τοποθεσιών, ε, οι οποίες μπορούν να γίνονται επισκέψιμες. 30 εκατομμύρια άτομα έλαβαν χώρα στις συναντήσεις που έγιναν ε, ε, αυτή τη χρονιά και είχαν την ευκαιρία να επανασύνδεθούν με την εθνική, τοπική και ευρωπαϊκή ταυτότητα. Στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, η το, το motive ήταν ε, η ε, κουλτούρα όσο παράγοντας ε, αξιοπρέπειας και ένωσης. Στη Βουλγαρία και το Λουξεμβούργο από την άλλη μεριά οι συναντήσεις έφεραν διπλάσιο κοινό από τα προηγούμενα χρόνια. Στην Σουηδία 250 εκδηλώσεις, περισσότερες από το 2017 διοργανώθηκαν φέτος και με τη συμμετοχή πολλών κοινοτήτων, πολιτικών κοινοτήτων, εθνοτικών κοινοτήτων, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την ανεκτικότητα και να καταπολεμήσουμε τη μυσαλλοδοξία. Ε, οι μέρες πολιτικής χρονομιάς προφανώς ήταν ε, πολύ σημαντικά γεγονότα, αλλά έλαβαν χώρα και άλλες εκδηλώσεις. Ε, άτομα αλλά και οικογένειες σε όλη την Ευρώπη είχαν την ευκαιρία να ε, επανερμηνεύσουν τη δική τους ταυτότητα. Η Europa Nostra, από την άλλη μεριά, κινητοποίησε όλους όσοι ενδιαφέρονται για την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης. Η Νέσκα θα μας πει περισσότερα για αυτά τα πράγματα σήμερα. Εξετάζοντας ε, τη σχέση ανάμεσα στην κουλτούρα, τον πολιτισμό και την ταυτότητα, πρέπει οπωσδήποτε ταυτόχρονα να προστατεύουμε και να συντηρούμε την πολιτική μας κληρονομία. Και αυτό μας φέρνει στο δεύτερο πάνελ. Η Σούζαν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συντηρητών Εργών θα μας μιλήσει αργότερα. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά φέτος ε, στο πλαίσιο της ε, Ευρωπαϊκής ημέρας συντηρητών στις 14 Οκτωβρίου. Η πολιτική κληρονομιά είναι σημαντική για την ταυτότητά μας, για το τι είμαστε και γι' αυτό λόγο θα πρέπει οπωσδήποτε να την προστατεύουμε. Στην προστασία αυτή είναι πολύ σημαντικό να περνάει κάθε φορά στην επόμενη γενιά η τεχνογνωσία που υπάρχει. Και η συντήρηση των, ε, της πολιτικής μας κληρονομιάς έχει ως στόχο να διατηρηθεί αυτή και ταυτόχρονα ε, να παραμείνει ακέραια. Σε όλη τη χρονιά δόθηκε έμφαση ειδικά σε αυτό. Ως παράδειγμα, η ομάδα εργασίας ε, εμπειρογνωμών σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάστηκε ε, κατευθύνσεις γραμμές ποιότητας για τη συντήρηση πολιτικής κληρονομιάς. Στην Βενετία θα παρουσιάσουμε αυτές τις... Ε, στη Βιέννη, συγγνώμη, θα παρουσιάσουμε αυτές τις κατευθύνσεις γραμμές. Και αυτές οι αρχέ το 2019 θα μπουν σε δημόσια διαβούλευση από την Κομισιόν έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν στην, ε, στις αποφάσεις που θα ληφθούν για τη χρήση ε, πόρων για τη χρηματοδότηση ε, της συντήρησης. Ε, είναι πολύ σημαντικό να συμμετάσχουν και οι κοινότητες που συμβιώνουν με την πολιτική κληρονομιά. Ένα project σχετικό ήταν οι πολιστικές διαδρομές. Οι διαδρομές αυτές ε, σκοπεύουν να ενώσουν ε, πόλεις στις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει ε, εκδηλώσεις για την πολιτική κληρονομιά. Αυτή η πρωτοβουλία συμπληρώνει την προσήλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια με την προοπτική της ένταξης. Μια πολιτική την οποία παρουσιάσαμε το Φεβρουάριο του 2018 ο τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, γνωρίζουμε ότι μπορεί από την άλλη μεριά να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης, αλλά θα πρέπει να λάβουμε μέτρα έτσι ώστε να είναι βιώσιμος. Βενετία, Ντουμπρόβνικ, Βαρκελόνη, τρεις πόλεις μεταξύ άλλων, ε, όπου οι κάτοικοι έχουν βγει στους δρόμους για να διαδηλώσουν κατά του υπερτουρισμού. Πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτή την πραγματικότητα. Μία από τις ε, δέκα πρωτοβουλίες του έτους ήταν ακριβώς η πρόθεση του βιώσιμου πολιστικού τουρισμού. Ε, καλωσορίζω τη δήλωση της Βαρκελώνας, καλύτερη, καλύτερη χώρη να ζούμε, καλύτερη χώρη να επισκεφτόμαστε, ε, τον ε, εμπλεκομένο στον τομέα του τουρισμού και της πολιτικής κληρονομιάς. Ε, αυτή η δήλωση προτείνει μια σειρά αρχών έτσι ώστε να εξισορροπήσουμε υπεύθυνα την διατήρηση της πολιτικής κληρονομιάς, τις απαιτήσει του τουρισμού και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Επιπλέον, άλλα σχέδια εστιάζουν στη σχέση ανάμεσα στη φυσική και την πολιτιστική κληρονομιά. Διαβάζω πάρα πολύ γρήγορα γιατί φοβάμαι το σφυρί της πέτρα. Οι υπηρεσίες ε, ε, οικοσυστημάτων του, της Natura 2000 έχουν τη δυνατότητα να εντείνουν αυτούς τους δεσμούς. Για παράδειγμα, η Actelec και η ε, οι ε, σπηλιές της ε, Σλοβακίας κοντά στη σύνορα με την Ουγγαρία. Εκεί προσπαθούν οι Σλοβάκοι να αναπτύξουν τον οικολογικό τουρισμό με παράλληλη διατήρηση των σπηλιών αλλά και της ε, φύσης και της πανίδας γύρω από αυτές. Εκεί καθορίζονται ζώνες για την άγρια φύση, περιοχές που ε, είναι επισκέψιμες μόνο μέσω συγκεκριμένων μονοπατιών και άλλες που είναι ελεύθερης επίσκεψης. Και οι τοπικές κοινότητες συμμετέχουν ε, έντονα και στενά ε, στην δημιουργία αυτού του οικολογικού βιώσιμου τουρισμού. Εξαιτίας ε, γεωγραφικών καταστροφών όμως ε, σημαντικά κομμάτια της κληρονομιάς μας μπορεί να καταστραφεί. Δυστυχώς όμως, ευτυχώς όμως καινούργιες τεχνολογίες μπορούν να μας βοηθήσουν ε, στην συντήρηση και την επισκευή πολιτικής χρονιά. 66 εκατομμύρια ευρώ διοχετεύθηκαν σήμερα για, την, για αυτό ακριβώς το θέμα. Η Κομισιόν, για παράδειγμα, χρηματοδότησε τέσσερα προγράμματα έρευνα και καινοτομία προκειμένου να δοκιμαστούν νέε λύσει για να διαχειριστούν οι ε, κίνδυνοι ε, που βαραίνουν την πολιτική κληρονομιά σε περιπτώσεις ε, φυσικών καταστροφών. Επίσης τεχνολογίες για να αξιολογούνται οι ζημιές που έχουν προκληθεί και να προγραμματίζεται η επισκευή τους. Επίσης, ένα ε, προχωρημένο, ε, μια προχωρημένη συσκευή λέιζερ, ε, κινητή συσκευή λέιζερ, που δημιουργεί σχέδια σε τρεις διαστάσεις που θα βοηθήσουν στο έργο των επιστημόνων. Για παράδειγμα, στη Βασιλική της Νότσια στην Ιταλία, που είχε πληγεί από τους σεισμούς. Και περνάω στο τελευταίο θέμα μου. Όλα αυτά δεν θα είχαν καμία σχέση αν δεν εστιάζαμε στην εκπαίδευση των νέων. Τι κάνουμε με τους νέους, πώς αποσπούμε το ενδιαφέρον τους, πώς τους εμπνέουμε. Όσο παρόλο ότι δεν έχουμε μια σαφή απάντηση αυτή τη στιγμή πρέπει σε εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο να κάνουμε την προσπάθεια. Θα πρέπει οι δάσκαλοι και οι καθηγητές να φέρουν την πολιτική κληρονομιά στην ε, αίθουσα διδασκαλίας. Ε, έχουμε ηλεκτρονικές διδημοποιήσεις, έχουμε ένα διδακτικό kit για το εκπαιδευτικό προσωπικό, ε, έχουμε ένα βιβλίο για τις ε, ηλεκτρονικές διδημοποιήσεις, με παραδείγματα για το πώς η πολιτική κληρονομιά μπορεί να ξαναέρθει στις τάξεις. Καλεί τους φοιτητέ και του μαθητέ να σκεφτούν αυτά τα θέματα μέσω της ε, πολιτιστικής έκφρασης, μέσω εκθέσεων, μέσω ανταλλαγών με άλλους μαθητές σε άλλες χώρες και σκεπτόμενοι για το τι είναι αυτό που μας ενώνει. 600.000 δάσκαλοι συμμετέχουν στις ε, ηλεκτρονικές δημοποίησεις, οπότε θα φτάσουμε σε ένα πολύ ευρύ κοινό. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ε, ε, φέρνει τους νέους σε επαφή με τους συντηρητές. Στο Erasmus Plus έχουμε την πολιτική κληρονομιά ως προτεραιότητα για όλες τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις και τελειώνω πρόεδρε. Ο Επίτροπος Ναύρασιτ θα σα πει ποια είναι τα σχέδιά του, έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό τη Πολιτική Κληρονομιάς να αφήσει μια κληρονομιά για το μέλλον. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον στις παρατηρήσεις του, είμαι σίγουρη. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Ja, vielen, vielen herzlichen... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέμης, ευρύτατη παρουσίαση για τις δραστηριότητε της ε, Κομισιόν και για την χρήση των ε, διαφορών προγραμμάτων για την πολιτιστική κληρονομιά και ευχαριστώ βεβαίως και την ε, Πρέσβη Confind για την πολύ καλή παρουσίαση που μας έκανε για το πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα της Αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου αυτό το τελευταίο εξάμεινο στα πλαίσια του πολιτιστικής κληρονομιάς και βεβαίως χαίρομαι που μπορώ να έρθω στην διάσκεψη την, ε, το Δεκέμβριο στη Βιέννη. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πρώτο πάνελ για να δούμε το θέμα της ε, ταυτότητας και του πολιτισμού. Ε, το πάνελ έγινε χτες, του οποίου προείδρευσε η κυρία Σίλβια Κώστα και θα ήθελα να της δώσω το λόγο για τρία λεπτά, ώστε σύντομα να μας παρουσιάσει τι διεμήφθη αυτό το πάνελ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Πρέσβυρα για τα λόγια της ε, και για την δέσμευση Ευχαριστώ την Γενική Διευθύντρια Χριστοφίδου, ε, την υποστήριξη της Επιτροπής ε, και τις πολλές προοπτικές που ανοίγονται. Ε, ευχαριστώ επίσης τους πολλούς συμμετέχοντες στο πρώτο πάνελ που ήταν εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων, ενδιαφερομένων φορέων και τριών γενικών διευθύνσεων. Ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας ε, ε, μιλώντας ακριβώς για την περιπλοκότητα της ε, ευρωπαϊκής ταυτότητας επί τη βάση της πεποίθησης ότι δεν υπάρχει καμία αντίφαση μεταξύ της διαφορετικότητας των εθνικών ταυτοτήτων και της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Και κινώντας ακριβώς από την πολλαπλή ταυτότητα, όπως και πολλοί ενδιαφέρουσες μελέτες εντόπισαν θα πρέπει ακριβώς επί της περιπλοκότητας αυτής να εστιαστούμε ώστε να βρούμε ένα κοινό παρελθόν και τις πολλαπλές ταυτότητες οι οποίες συνθέτουν το ευρωπαϊκό πρόσωπο, τις εθνικές ταυτότητες. Ε, σκέφτομαι τον ε, Λεωνάρντο Νταβίντσι που ήταν Ιταλός, το Σκάνος και βεβαίως Ευρωπαίος. Ε, μπορούμε λοιπόν από κοινού να δημιουργήσουμε μια σύνθετη εικόνα, ένα παλίμψιστο από αυτές τις ταυτότητες ε, που συνθέτουν τη σημερινή Ευρώπη. Και γι' αυτό και τα προγράμματα των εθνικών σχολείων είναι πάρα πολύ σημαντικά επ' αυτού και ενώνουν το παρελθόν μας με το κοινό μας μέλλον. Οι φετινές πρωτοβουλίες ε, δημιουργούν και μια κοινότητα από την εκδήλωση στο Μιλάνο μέχρι τη σύνοδο την πολύ σημαντική στο Βερολίνο δημιουργείται αυτή η Heritage Community μαζί με την ε, σύμβαση του Φάρο που καλό πολλές ε, χώρες να επικυρώσουν. Ε, αναδύεται λοιπόν μια εικόνα πολλαπλών κέντρων της Ευρώπης και πρέπει να βασιστούμε από αυτά τα κέντρα για να καταλάβουμε την σύνθετη ταυτότητα της Ευρώπης. Για παράδειγμα, η 21η Σεπτεμβρίου και οι καμπάνες που ηχούσαν σε όλη την Ευρώπη. Όλα αυτά ε, συνθέτουν ε, και σε μια ε, ψυχική, ψυχολογική διάσταση, γιατί δεν πρέπει μόνο διανοητικά να κατανοούμε αυτά τα πράγματα, να τα προσεγγίζουμε, αλλά και συναισθηματικά. Προέκυψαν πολλές απαντήσεις από τη συζήτηση του πάνελ, αλλά και πολλά ερωτήματα. Πρέπει να οικοδομήσουμε γέφυρες μεταξύ των διαφόρων ταυτοτήτων, εθνικών, τοπικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών και πρέπει να μιλούμε για, την, ε, για το κληροδότημα και το θρησκευτικό εκτός του πολιτιστικού που ενώνει όλους εμάς ως Ευρωπαίους. Επομένως είναι απτά αλλά και μία απτά στοιχεία που προκύπτουν ε, ως ε, θεμελιώδη συστατικά αυτής της ταυτότητας η Σουηδή συνάδελφος ε, προβληματίστηκε σχετικά με ε, τους όρους, ε, τους εθνικιστικούς που χρησιμοποιούνται καμιά φορά για να θυμίσουν αυτήν την ταυτότητα την ευρωπαϊκή. Βεβαίως έχουμε και μια κοσμική παράδοση που βασίζεται σε μια ολόκληρη ιστορία φιλοσοφίας, ιστορίας κτλ. Ε, το έτος το αφιερωμένο ε, ήταν και το εφαλτήριο για πάρα πολλά έργα, πάρα πολλά προγράμματα υπό την ε, γραμμή Δημιουργική Ευρώπη. Θα κλείσω αμέσως επί τελευταίων δύο σημείων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η εκπρόσωπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μίλησε για μια, ένα μοντέλο διακυβέρνησης πολυεπίπεδο ε, και γέφυρες μεταξύ των γενεών που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και νομίζω ότι στο σχέδιο δράσεως θα πρέπει αυτό να ενισχυθεί. Οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, τόνισαν ότι η ταυτότητα ευρωπαϊκή είναι μια διαδικασία και όχι ένας ε, καθεαυτός αυθύπαρκτος στόχος. Η σύνδεση επίσης της εκπαίδευσης με την πολιστική κληρονομιά συνθέτει προς την επίτευξη μιας ε, σύνθετης ταυτότητας και πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας ώστε και στις υποψήφιες χώρες που έχουν ζήσει συγκρούσεις πολεμικές και σημαντικές δυσκολίες θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως καταλήτης και κλείνω με μια φράση που ήδη αναφέρθηκε, μου φαίνεται πολύ σημαντική. Το ευρωπαϊκό έτος της πολιτιστικής κληρονομιάς ήταν υπερβολικά σύντομο για να μην γίνει υπερβολικά μεγάλο. Είναι μια φράση που ήθελα να την αναφέρω γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας, για το τι έγινε στην χθεσινή συνάντηση. Να δούμε λοιπόν τους ομιλητές για το πάνελ πολιτισμός και ταυτότητα. Ξεκινούμε με την Σνέσκα Κβάτφλικ Μιχαήλοβιτς, γενική ε, γραμματέα της Europa Nostra. Ε, πέντε λεπτά με την ε, προϋπόθεση ότι μπορείτε και να μην τα χρησιμοποιήσετε όλα. Σας ακούμε. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Εθνικών Κοινοβουλίων, αγαπητοί φίλοι, είναι τιμή και ευθύνη για μένα που είμαι η φωνή της κοινωνίας των πολιτών σε αυτήν τη συνάντηση που συνενώνει μέλη των κοινοβουλίων και μέλη ενδιαφερομένων φορέων για να συζητήσουμε το κληροδότημα του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς και γιατί είναι τόσο ιστορικό αυτό το έτος. Όχι μόνο γιατί είναι το μόνο θεματικό έτος υπό την Επιτροπή Juncker, αλλά είναι το πρώτο έτος που ξεκίνησε από κάτω προς τα πάνω ξεκίνησε από τους ενδιαφερομένους φορείς εθνικά και ευρωπαϊκά. Και ευτυχώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αγκάλιασε την ιδέα αυτή και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο ώστε να πείσει τον πρόεδρο Γιούνκερ ότι αυτή η ιδέα άξιζε να την υποστηρίξουμε. Στην ανάμνηση των 100 ετών του τέλους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου πρέπει να θυμόμαστε και να μην ξεχνούμε ποτέ ότι είναι ειρηνική η στόχευση και το όραμα εδώ. Πρέπει να θυμόμαστε τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και το γεγονός ότι πάντα μας οδηγούν οι αξίες και οι αρχές μας. Είναι σημαντικό να θυμίζουμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα είναι και πολιτιστικό βεβαίως. Απέναντι σε τόσες πολλές προκλήσεις αλλά και απειλές ακόμα απέναντι στις βασικές μας αξίες πρέπει να αλλάξουμε το ύφος, να αλλάξουμε το αφήγημα σχετικά με την Ευρώπη. Έχουμε μια πλούσια κληρονομιά ηλική και μη, έχουμε κοινή ταυτότητα, κοινή ανάμνηση, κοινή προέλευση. Είμαστε προϊόντα ανταλλαγής αιώνων, όχι μόνο μεταξύ καλλιτεχνών και επιστημόνων, αλλά και κοινών ανθρώπων και κοινοτήτων, κοινωνιών. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε περισσότερο με το ευρωπαϊκό όνειρο, θα πρέπει να ενισχύσουμε μια αίσθηση κοινή ταυτότητας κοινού ανήκειν και όπως είπε και η κυρία Κώστα, αυτό έχει πολλαπλά επίπεδα, είναι σύνθετο. Αυτά τα επίπεδα δεν ανταγωνίζεται το ένα το άλλο, αλλά συνθέτουν μια συνολική εικόνα. Κάθε ιστορικό μνημείο, κάθε αρχαιολογικός χώρος, καλλιτεχνικός χώρος μας ε, αφηγείται μια ιστορία τοπική αλλά και ευρωπαϊκή και όλοι μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για την εθνική μας, τοπική μας ταυτότητα αλλά και για την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα. Και αυτό είναι το μήνυμα του έτου. Εχθές είχαμε ένα workshop υπό την προεδρία της κυρίας Κώστα ε, στον οίκο της ευρωπαϊκής ιστορίας που ήταν συμβολικό. Αναφερόμαστε στην παιδεία, στην εξιστόρηση, δηλαδή στην διδαχή της ιστορίας, χωρίς την οποία οι τωρινέ και μελλοντικέ γενιές δεν θα είναι σε θέση να κατανοήσουν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα και δίνοντας έμφαση στην διδαχή της ιστορίας πρέπει να έχουμε πολλαπλά οπτικά σημεία, πολλαπλές προοπτικές, ώστε οι νέοι άνθρωποι να έχουν καλύτερα, περισσότερα μέσα να είναι Ευρωπαίοι πολίτες, να ανθίστανται σε λαϊκιστικές ή εθνικιστικές αφηγήσεις, λέει ο Μιλήτρια, σχετικά με ιστορικά γεγονότα. Αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, αυτό το ευρωϊκό έτος ήταν η χρυσή ευκαιρία για να αναγνωρίσουμε τα πολλαπλά ωφέλη της κοινή μας παράδοσης για τις κοινωνίες, την οικονομία, το περιβάλλον μας και την κοινή μας ταυτότητα, αλλά και για να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές απειλές προς όλα αυτά. Ενισχύσαμε τις ε, παρούσες συμμαχίες, δημιουργήσαμε καινούργιες, είχαμε ένα πολύ σημαντικό σημείο καμπής του mainstreaming της ιστορικής ε, πολιτιστικής μας κληρονομιάς μέσα στα προγράμματα, τα εκπαιδευτικά και τα των πολιτικών μας. Θα ήθελα να κλείσω αναφερόμενη ε, στο, στην επίκληση για δράση τον περασμένο Ιούνιο στην Σύνοδο του Βερολίνου η Ευρώπα Νόστρια είχε την τιμή να συνδιοργανώσει μαζί με την Γερμανική Επιτροπή μας τον συντονιστή δηλαδή στη Γερμανία, είπαμε ότι η ώρα για δράση είναι τώρα. Καλούμε για ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την πολιτική κληρονομιά και είμαστε πανευτυχείς που η Επίτροπος θα παρουσιάσει στη Βιέννη το σχετικό πρόγραμμα. Και μάλιστα είχαμε και το συμβολικό μέγεθος 2018 υπογραφές, μεταξύ των οποίων η κυρία Κώστα ε, ε, ο Μριτσέα και άλλοι, θα ήθελα αυτό να διαβαστεί ως μήνυμα σε όλα τα κοινοβούλια, στις ενώσεις, ε, στους φορείς. Αλλά όπως είπαν και οι συνάδελφοι, 11 μήνες είναι υπερβολικά βραχή διάστημα για μια τέτοια προσπάθεια. Έχουμε την κοινή ευθύνη, οι πολιτικοί ηγέτες, οι υπεύθυνοι των ενδιαφερομένων φορέων και των ενώσεων, να δημιουργήσουμε την ε, ισχύ της κοινή μας ταυτότητας για να δώσουμε ένα βαθύτερο νόημα και κατεύθυνση σε όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Σνέσκα. Πάμε τώρα να ακούσουμε την Μαργαρίδα Μάνο. Είναι μέλος της Πορτογαλικής Βουλής. Σας ακούμε για πέντε λεπτά. Συγχαρητήρια στην κυρία Πρόεδρο. Ε, καλωσορίζω και χαιρετίζω όλους και όλες. Στην... Ενωμένη στην ποικιλομορφία είναι το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σύνθημά της. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση χωρών που θέλουν να εργαστούν για την ειρήνη και χαρακτηρίζεται από μια ποικιλομορφία πολιτισμών, γλωσσών κλπ. Μια κοινωνία η οποία είναι ενωμένη μέσω της ποικιλομορφία, όπου η ποικιλομορφία επιτρέπει μια πιο πλούσια Ευρώπη. Αυτή είναι η πρόκληση που βασίζεται στην πολυφωνία των πολιτισμών, των παραδόσεων και των γλωσσών. Η συμβιωτική σχέση ανάμεσα στον πολιτισμό και τη γλώσσα είναι πολύ γνωστή και ορίζεται ως ένα συμβολικό σύστημα που ε, έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει αξίες ε, ε, και ταυτότητες μέσω του διαλόγου. Οπότε η γλώσσα δημιουργεί ένα χώρο που μοιράζεται. Μια, χώρα με 24, μια Ευρώπη με 24 επίσημες γλώσσες και πάνω από 60 τοπικές σημειωτικές γλώσσες είναι ένας πολιτιστικός θησαυρό. Ένας τεράστιος ε, χώρος ε, που, όπου μοιράζονται αξίε και μέλλον. Είναι ο λόγος ύπαρξης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η πολιτική λοιπόν της ε, πολυγλωσσίας θα πρέπει να ενταθεί προς δύο κατευθύνσεις. Η προστασία της γλωσσικής ποικιλομορφίας στην Ευρώπη και η πρόθεση της εκμάθησης γλωσσών. Ε, δεν αυταπατώμεθα. Ε, το μέλλον δεν θα είναι μόνο γλωσσικό όπως κάποιοι πιστεύουν στην κοινωνία της γνώσης. Η γλώσσα είναι μια έκφραση της γνώσης ε, που έχει μεγάλη ποικιλομορφία και κάθε γλώσσα έχει το δικό της ε, πλούτο που επιτρέπει να περάσει μέσω αυτής ένας ολόκληρος πολιτισμός. Η πολιστική πυγρομορφία λοιπόν είναι ποικιλομορφία και στη γνώση και αντιπροσωπεύει μια στρατηγική αξία που ε, υποχρεώνει την Ευρώπη να ε, δημιουργήσει, να φροντίσει όλες τις γλώσσες, τις περιφερειακές, τις ε, και τις εθνικές. Ε, ανήκοντας στην Ευρώπη ανήκει κανείς στον κόσμο. Ε, η πορτογαλική γλώσσα μιλιέται από 10 εκατομμύρια Πορτογάλων αλλά και 250 εκατομμύρια σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Τα πορτογαλικά είναι γλώσσα πιο πολύ μιλιέται στο νότιο ημισφαίριο με 217 εκατομμύρια άτομα που τη μιλούν. Είναι η έκτη γλώσσα που πιο πολύ μιλιάται σε όλο τον κόσμο, πέμπτη στο ίντερνετ, τρίτη στα, δίκτυα, στα, ε, στα ε, μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Twitter. Ε, με αυτή τη διάσταση που έχει μπορεί να ανοίξει την Ευρώπη σε όλο τον κόσμο, στον πραγματικό και τον ψηφιακό κόσμο, όπου μπορεί να προκύψει μια απτή πραγματικότητα, μια ένας πολιτισμός που θα είναι παρόν σε όλο τον κόσμο. Η ενίσχυση της ταυτότητας Ευρώπης ε, δεν μπορεί να αγνοεί μια ε, δυναμική πολιτική προστασία της πολιτικής και της γλωσσικής κληρονομιάς. Ο δεύτερος άξονας έχει σχέση με την εκπαίδευση και την εκμάθηση γλωσσών. Η Ευρώπη έχει ως ευγενή στόχο κάθε Ευρωπαίος να μιλάει τη γλώσσα του και άλλες δύο τουλάχιστον γλώσσες. Ο καλύτερος τρόπος να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι η το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα να περιλαμβάνει δύο ξένες γλώσσες. Η γνώση ξένων γλωσσών δημιουργεί, βελτιώνει το διάλογο, την αλληλοκατανόηση, ε, την ανάπτυξη οικονομική και κοινωνική, καθώς επίσης ε, βελτιώνει και τη συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή το 80% των μειονοτικών γλωσσών της Ευρώπης διατρέχουν κίνδυνο εξαφάνισης, οπότε χρειάζεται η εκπαίδευση και σε αυτές τι γλώσσε. Ο Φερνάντο Πεσόα, ο πιο παγκόσμιο πορτογαλο ποιητή, το πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα, ήξερε αρκετέ άλλε γλώσσε. τα αγγλικά, τα ισπανικά, τα γερμανικά, ακόμα και τα λατινικά και τα αρχαία ελληνικά. Ε, και στο, λίβρο, στο βιβλίο τη ανησυχία, έγραψε ε, «Πατρίδα μου είναι η πορτογαλική γλώσσα». Ο Εντουάρντο Λορένσο, φιλόσοφος, και ε, θαυμαστής του Πεσόα έγραψε «Μια γλώσσα δεν ανοίξε κάποιον συγκεκριμένο, αλλά και εμείς δεν είμαστε τίποτα χωρίς, ε, ε, αν δεν κάνουμε τη γλώσσα δική μας. Στην Ευρώπη ε, δεν θα έχουμε ταυτότητα ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, αν δεν είναι δικές μας περισσότερες από μία γλώσσες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σα Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφε, που μας μιλήσατε και για την αξία της γλώσσας στην ε, ευρωπαϊκή ταυτότητα. Και ε, τώρα ασχολούμαστε μάλιστα και με μια πρόταση της, ε, μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακριβώς για τις για το πώς μπορεί κανείς να μάθει γρήγορα και αποτελεσματικά δύο γλώσσες τουλάχιστον και ελπίζω ότι και τα κράτη-μέλη θα κάνουν βήματα ως προς αυτό. Πάμε τώρα στον, στην επόμενη ε, ομιλήτρια, η Καμέλια Γκραβίλα από την Ρουμανική Βουλή. Πού βρίσκεται? Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Uh, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας παραθέσω κάποιες σκέψεις για, τον, για την εκπαίδευση, τις διαπολιτισμικές προσεγγίσεις. Βρισκόμαστε στο τέλος σε μια σημαντική χρονιά, σε μια χρονιά που είναι συμβολική, που περιείχε πολλές δράσεις. Μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτές τις αξίες και από φιλοσοφική και από παιδαγωγική σκοπιά και βεβαίως πρέπει να ξεκινήσουμε με το σκεπτικό ότι ο πολιτισμός είναι ένα κομμάτι μας, ότι ανήκουμε σε έναν κόσμο, σε μια χώρα, με μια ιστορία, με μια συγκεκριμένη γεωγραφία. Ζούμε με συγκεκριμένε αξίες και αρχές. Ελπίζω ότι βλέπετε τις ε, διαφάνειες ε, που παρουσιάζουν τις ε, ιδέες μου. Η ε, εκπαίδευση, η θρησκεία, η τέχνη, οι πνευματικές αρχές είναι ε, οι αρχές ακριβώς που διέπουν την, ε, το πνευματικό μάτριξ στο οποίο ανήκουμε. Βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι σε έναν διεθνή κόσμο δεν μπορούμε να ζούμε σε μόνο πολιτιστικούς κόσμους. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους νέους μας να δεχτούν την πολυπολιτισμικότητα, να δέχονται και να κατανοούν τη διαφορετικότητα και να προσαρμόζονται όσο πιο γρήγορα γίνεται στον καινούριο αυτό κόσμο. Και επίση το πρόβλημα είναι με του ε, ενήλικε. Για αυτού ίσω είναι πιο δύσκολο γιατί έχουν σαφεί, εδρεωμένε πεπιθήσει. Οπότε πρέπει να μιλήσουμε σε πολύ παραδοσιακέ κοινωνίε, σε πολύ συντηρητικέ κοινωνίε. Και υπάρχει κι άλλο ένα κίνδυνο. Ε, η διαπολιτισμική ανισορροπία, που, όπως το ονομάζουν οι ανθρωπολόγοι. Γιατί ζει κανείς μεταξύ δύο πολιτισμών ή περισσότερων πολιτισμών. Έχεις τις δικές σου ιδέες, τις δικές σου αξίες και θέλεις να ε, εκτιμώνται από τους άλλους. Αλλά από την άλλη πρέπει να κατανοήσεις και εσύ ότι πρέπει να είσαι δεκτικός και ευαίσθητο απέναντι σε άλλες κουλτούρες. Η μόνη λοιπόν λύση και η μόνη λογική, ιδεολογική επιλογή σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι να εκπαιδεύσουμε μέσω αυτή τη διαπολιτισμική προσέγγιση τους πολίτες και να καταλάβουμε ότι έχουμε μια βάση πολιτιστική, εθνική, ταυτότητα και μπορεί να είναι αυτή η δική μας προσωπική ταυτότητα, η τοπική, η εθνική μας ταυτότητα, αλλά έχουμε και την διεθνή πτυχή και πρέπει να μπορούμε αυτό να το κατανοήσουμε. Πώς το κάνουμε αυτό, μέσω προγραμμάτων, μέσω ανταλλαγών, μέσω εκπαίδευσης, μέσω γνώσης κτλ. Και πρέπει να σκεφτούμε και την επίσημη άτυπη ε, εκπαίδευση, όχι μόνο της εντυκλίους, εμείς ως εκπαιδευτικοί επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ σε εξετάσεις, σε εγκυκλίους, ακαδημαϊκές και ξεχνούμε ότι πρέπει να διαμορφώσουμε προσωπικότητες, να εκπαιδεύσουμε τους πολίτες που θα ζήσουν σε πολύ διαφορετικές κοινωνίες από τις δικές μας. Και πρέπει επίσης να καταλάβουμε ότι οι φοιτητέ μας, οι σπουδαστέ μας πρέπει να έχουν κατανόηση και να είναι ανοιχτοί στην διαφορετικότητα. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί, ας σκεφτούμε πώς είναι δομημένα τα εκπαιδευτικά συστήματα στις χώρες μας και πώς μπορούν αυτά να προετοιμάσουν τους φοιτητέ για να συναντήσουν τον άλλον, τον διαφορετικό και πώς μπορούν να τον αποδεχτούν. Η ε, απάντηση είναι διαφορετική βεβαίω ανά χώρα και γι' αυτό χρειάζονται κάποιες κοινέ αρχές, αξίες, κατανόηση, ανοιχτικότητα, ανοιχτό πνεύμα και αν το δούμε και από φιλοσοφική σκοπιά ή ανθρωπολογική σκοπιά, οι μεταμοντέρνε κοινωνίες είναι ένα παγκόσμιο χωριό, ένα τεχνικός κόσμος, ένα παζλ μικρών συμπάντων. Και η υποχρέωσή μας ως εκπαιδευτικών ή πολιτικών είναι να βρούμε μια συνεκτικότητα, μια συνοχή μεταξύ όλων αυτών των πτυχών. Από την ε, λογοτεχνία, από την εκπαίδευση, μέχρι να μπορέσουμε να κατονοήσουμε το τι συμβαίνει στον κόσμο. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Αυτό που θέλω εγώ να υπογραμμίσω στο τέλο τη παρέμβασή μου είναι ότι οι, οι πολιτισμικές, ε, τα διαπολιτισμικά προσόντα, η κατανόηση, οι ανταλλαγέ, οι εκπαιδευτικέ επισκέψει, η φιλοσοφική κατανόηση τη προόδου είναι οι μόνε λύσει μέσω των οποίων οι φοιτητέ, οι νέοι και οι μεγαλύτεροι μπορούν να κατανοήσουν το διαφορετικό. Είναι σημαντικό και στι εθνικέ εγκυκλίου, είτε μέσω λογοτεχνία, είτε μέσω ε, ε ξένη λογοτεχνία, ε, κοινωνικών επιστημών, θα πρέπει να υπάρχει αυτή η διαπολιτισμική προσέγγιση ως υποχρεωτικό μάθημα. Ίσως να είναι υπερβολικό αυτό που λέω, αλλά πρέπει να γίνει. Σε κάθε εκπαιδευτικό σύστημα θα μπορούσε να γίνει. Τέλος, Είμαστε ένα μέλος της ε, Ευρωπαϊκής Υπήρου, ανήκουμε σε αυτή την κοινή πολιτιστική κληρονομιά, αυτή είναι που μας ενώνει και είναι σημαντικό αυτό να μπορέσουμε να το κατανοήσουμε. Και να κατανοήσουμε βεβαίως ότι το να περιορίζουμε τους πολιτισμούς και να ζούμε μόνο μέσα στο δικό μας μα κάνει πιο φτωχού γιατί δεν καταλαβαίνουμε την ομορφιά τη ευρωπαϊκής κληρονομιάς, ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Ε, νομίζω ότι καταλάβαμε όλοι ότι μιλήσατε από την καρδιά σας. Ε, χαίρομαι πολύ που δεν ε, παίρνουν μόνο μέλο εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων στη διάσκεψη αυτή, αλλά σχεδόν όλε οι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων εκπροσωπούνται σήμερα εδώ, με του δικού του εκπροσώπου από τα κοινοβούλια του δεν είστε ακόμη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η παρουσία σας πραγματικά δείχνει ότι συνδεόμαστε όλοι στενά και γι' αυτό χαίρομαι πολύ που μπορώ να καλωσορίσω την Τραγκάνα Κώστης από το Σερβικό Κοινοβούλιο για να την ακούσουμε. Πού είναι? Ωραία, σας ακούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε ε, αγαπητοί φίλοι, αγαπητά μέλη των Εθνικών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχω την τιμή να σας μιλώ εκπροσωπώντας την Δημοκρατία της Σερβίας με αυτή την πολύ σημαντική για εμάς συνάντηση. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με τα ε, λόγια του Στέπαν Νέμανιε του 12ου αιώνα «Προστατεύστε την παράδοσή σας σαν τη ζωή σας» γιατί ένας ε, λαός που θα έχει, χαλέσει, που θα έχει απολέσει τη γλώσσα του, θα έχει απολέσει τη μνήμη του. Και γι' αυτό σας μιλώ σήμερα στη μητρική μου γλώσσα, για τι απειλέ που αντιμετωπίζουμε ως ταυτότητα σερβική και σε κάτι που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως πολιτισμική γενοκτονία. Αυτό το βλέπουμε στις, ε, την, Μάλλον η ταυτότητα αυτή απεικονίζεται στην Κρατσανίτσα, στην παλαιότερη από τις εκκλησίες που έχουμε από τον 4ο αιώνα και πολλές, πολλά σημαντικά μνημεία και εκκλησίες στο μετόχι και το κοσυφοπέδιο που είναι εγγεγραμμένα στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO ως απειλούμενα μνημεία και αυτό έχει συγκεκριμένη αιτία ένα τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς της Σερβικής σημαντικές τοιχογραφίες επίσης που έχουν αποσταλεί μέσω ε, δορυφορικού σήματος προς το σύμπαν ως ε, εκπροσωπώντας ε, την ανθρωπότητα. Τα μνημεία λοιπόν της πολιτιστικής κληρονομιάς σηματοδοτούν την ε, μερικές ώρες μαρτυρική πορεία του σερβικού λαού της, ε, το πάθος του σερβικού λαού μέσω των πολέμων του πρώτου παγκοσμίου πολέμου μεταξύ άλλων τα πολλά θύματα που είχαμε στους διάφορους πολέμους οι κατακτητές που ήταν πολυάριθμοι δυστυχώς ε, γενικώ στα Βαλκάνια και πέρασαν από τη χώρα μας, το βομβαρδισμό του Βελιγραδίου από τις ε, γερμανικές δυνάμεις ε, το 1941, όπου ένα από τα πρώτα θύματα του βομβαρδισμού αυτού ήταν η βιβλιοθήκη στο Βελιγράδι, ανεκτήμη της πολιτιστικής αξίας. Αυτή λοιπόν η πολιτιστική γενοκτονία είναι αυτή στην οποία αναφερόμουν νωρίτερα και οι απειλές προς την ε, πολιτιστική μας ταυτότητα με την καταστροφή βιβλίων αρχαίων μεσαιωνικών από τα πρώτα βασίλεια της Σερβίας ε, μαρτυρίες από την τουρκική ε, κατάκτηση και από την απελευθέρωση. Δυστυχώς σήμερα αυτές οι δράσεις ε, γίνονται υπό τα φώτα της διεθνούς κοινότητας ε, με διωγμό ε, Σέρβων από το κοσυφοπέδιο με καταστροφή των κατοικιών τους και ιστορικών νημείων και από την έλευση της διεθνούς ε, κοινότητας από το 1999 στην περιοχή 150 ε, ε, μοναστήρια και εκκλησίες έχουν καταστραφεί και χιλιάδες χιλιάδων αγιογραφίες που έχουν ακλαπεί και έχουν τεθεί σε λαθρεμπόριο. Αυτά είναι τα μνημεία, τα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς τα οποία απειλούνται και καταστρέφονται στο κοσυφοπέδιο. Οι διεθνείς δυνάμεις ε, κατέγραψαν πως το 2004 κατέστρεψαν άλλα 26 μοναστήρια ε, και εκκλησίες στη Σερβία. Κανείς δεν θεωρήθηκε υπεύθυνο για τις πράξεις αυτές. Επομένως ε, πρόκειται για οργανωμένη επίθεση για να εξαφανιστούν τα ίχνη της ε, σερβικής ε, κληρονομιάς και ιστορίας από την περιοχή του Κωσυφοπεδίου. Και αυτό γίνεται με έναν πολύ πιο έμεσο τρόπο. Έχουμε δει ιστορική πλαστογράφηση στα τελευταία χρόνια άνευ όπου παρουσιάζονται ε, ιστορικές φυσιογνωμίες και ηγέτες της Εκκλησίας του Μεσαίωνα ως αλβανικής καταγωγής. Νομίζω ότι αυτικές, ε, αυτές οι απειλές έχουν, είναι άνευ προηγουμένου, είναι απολύτως οργανωμένες και νομίζω ότι η απειλή είναι απολύτως Ε, ε, αποδεδειγμένη και είναι και ένα στοιχείο πραγματικά ε, που θα έπρεπε να προκαλεί όνειδος στη διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα στα διεθνή, στους διεθνείς οργανισμούς που καλούν ότι η πολιτική... Διακόπτει η Πρόεδρος και ευχαριστεί την ομιλήτρια. Δυστυχώς πρέπει να είμαι αυστηρή γιατί αλλιώς δεν θα προλάβουμε. Λοιπόν, να χαιρετήσω τώρα τον πρόεδρο της ε, Επιτροπής ε, Πολιτισμού της Ισπανικής ε, Βουλής, Αλμπέρτο Γκουτιέρες Αλμπέρκα. Και τον καλό να πάρει το λόγο. Σας ακούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παίρνω το λόγο εκ μέρους της Ισπανικής Βουλής. Ορισμένοι πιστεύουν ότι η πολιτική, η πολιτική ταυτότητα δεν υπάρχει καν. Είναι περίπλοκο, αλλά εγώ πιστεύω ότι υπάρχει. Το θέμα είναι όμως και πώς κατασκευάζεται, πώς οικοδομείται η ταυτότητα, γιατί η δημιουργία μιας ταυτότητας σε αντίθεση με κάποιον άλλον, σε σύγκρουση με μια άλλη, μια ταυτότητα που βασίζεται στο φόβο, μερικές φορές μας στέλνει προς τη λάθος κατεύθυνση για τις ε, αξίες οι οποίες ε, στηρίζουν την ταυτότητα. Χτε συζητήσαμε το θέμα της οικοδόμηση, μια υπερεθνικής ταυτότητα που ξεπερνάει τι γλώσσε η οποία που, μια τέτοια ταυτότητα όμω που βασίζεται στι συγκρούσει ε, είναι ποδοσφαιρική. Ε, Θυμάμαστε εμεί πολύ καλά στην Ισπανία πότε κερδίσαμε το Ευρωπαϊκό Κύπελο Ποδοσφαίρου γιατί αυτή η νίκη δημιούργησε μια σημαντική ε, προσωρινή ταυτότητα, εθνική ταυτότητα πιο ισχυρή. Όταν περάσει όμως αυτή η εποχή ξεχνιέται αυτή η ταυτότητα. Οπότε ε, ε, οι χώρες όπως η Ισπανία που ερχόμασταν από αυταρχικά καθεστώτα ε, πλησίασαν ε, πολύ την ε, Ευρώπη γιατί αντιπροσώπευε τη δημοκρατία, την ελευθερία, τις, τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Και αυτή είναι η ταυτότητα την οποία επιθυμούμε. Ίσως θα έπρεπε αυτό το σύμφωνο που μας ενώνει να το τονίσουμε. Είναι οι αξίες τις οποίες μοιραζόμαστε και θα πρέπει να ξαναπλησιάσουμε την ευρωπαϊκή ταυτότητα με νέες αξίες όπως για παράδειγμα η ειρήνη, η οικολογία, η πρόσβαση σε αξιοπρεπείς μισθούς, ο σεβασμός της ε, γυναίκα, στη γυναίκα, η καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτές είναι πλέον οι αξίες της δύση που δημιουργούν ένα κοινό όραμα και μια καινούργια πολιστική ταυτότητα. Οπότε η αυτό το ευρωπαϊκό σύμφωνο ταυτότητας θα πρέπει να ανανεωθεί έτσι ώστε και οι καινούργιες γενιές να αντιμετωπίσουν την Ευρώπη ως ένα αξιόλογο ε, όραμα. Και, δεν θα, και αν το σχέδιό σου, το όραμά σου είναι ισχυρό, δεν φοβάσαι τις ταυτότητες, τις διαφορετικές ταυτότητες οικοδόμηση της Ευρώπης πάνω σε οικονομικές αξίες ε, των ταμείων συνοχής του κλπ. κλπ. Ε, δεν ακουμπάει, δεν αγγίζει τα αισθήματα των ανθρώπων. Γι' αυτό το λόγο είναι, σημαντική και, είναι σημαντικός και ο πολιτισμός. Εμείς μέσω του πολιτισμού ε, δημιουργούμε συναισθηματικές αξίες ο πολιτισμός είναι αυτός ο οποίος έχει δημιουργήσει την ταυτότητά μας. Για παράδειγμα, το Καμίνο Δε Σαντιάγο είναι μια διαδρομή προσκυνητών ε, πολλών αιώνων. Όμως έχει μετατραπεί πλέον σε μια πολιτιστική αξία ένωσης της Ευρώπης, διότι είναι πολλοί Ευρωπαίοι που επισκέπτονται, που κάνουν αυτή τη διαδρομή, αλλά είναι ταυτόχρονα και μια διαδρομή οικολογίας. Ε, είναι μια διαδρομή φιλοξενίας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πανδοχεία τα οποία φιλοξενούν τους προσκυνητές. Οπότε η πολιτική ταυτότητα δεν είναι μόνο μια ταυτότητα σφραγίδων. Ε, ακόμα και, στη, στο δρόμο του Σαντιάγο ε, οι προσκυνητές ε, παίρνουν σφραγίδες αναλόγω το που έχουν, από που έχουν περάσει, αλλά δεν αρκούν οι σφραγίδες. Η οικοδόμηση θα πρέπει να γίνεται μέσω της βιωσιμότητας, μέσω της βιώσιμης διαχείρισης του πολιτισμού και της, ε, και, και, ε, της φύσης. Έχει δοθεί το παράδειγμα της Βαρκελόνης, αλλά εγώ θα σας δώσω το παράδειγμα της Αλάμπρα, που είναι ένα παράδειγμα βιωσιμότητας. Συνεπώς θα πρέπει να εργαστούμε περισσότερο στο θέμα της βιωσιμότητας και από την άλλη μεριά στο θέμα της ψηφιακής κουλτούρας, του ψηφιακού πολιτισμού, γιατί ο ψηφιακός πολιτισμός μας δίνει το δρόμο για το μέλλον. τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να στηριχθούν και με τη χρήση τεχνολογιών και να περιλαμβάνουν και το ψηφιακό περιεχόμενο. Η ψυχή μπορεί να είναι κοινή, αλλά η ευφυΐα είναι κοσμοπολίτικη, είπε κάποιος. Και η πολιτική θα πρέπει να διέπεται από τον πολιτισμό, όχι από την οικονομία. Ε, όπως λέει οι Αμερικάνοι, οι Αμερικάνοι λένε είναι η οικονομία χαμένη, ε, τελικά είναι ο πολιτισμός χαμένε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Πάμε τώρα στην συζήτηση. Μέχρι στιγμής έχω εννέα ομιλητές για αυτό το πρώτο πάνελ. Έχουμε έξι λεπτά χρόνο. Άρα θα σας δώσω ένα λεπτό στον καθένα. Αλλά θα μπορούσα να προτείνω ε, όποιος από σας θέλει να πάρει το λόγο στο δεύτερο πάνελ, αν μπορεί. Γιατί στο δεύτερο πάνελ δεν έχουμε ακόμη μέχρι στιγμή ε, πολλού που να ζητούν το λόγο. Οπότε θα μπορούσατε ίσω να πάρετε το λόγο στον δεύτερο γύρο. Λοιπόν, ξεκινούμε τώρα. Πρώτος, ο Αρούνας Γκυλούνας, από τη Λιθουανία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Sorry. Uh, thank you, συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι, είναι πιεστικό το ένα λεπτό. Κυρίε και κύριοι, πρέπει να ομολογήσω ότι μερικέ φορέ ε, έχω την αίσθηση ότι ονειρεύομαι. Ότι δεν μιλούμε για την οικονομία, για την ασφάλεια, ούτε καν για πλαστικές σακούλες, αλλά για τον πολιτισμό. Εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ την κυρία Κώστα για την ε, για τον θαυμάσιο συντονισμό της ε, συζήτησης εχθές ε, και για την έκθεση. Εγώ πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Εμείς ε, γιορτάζουμε τα 100 χρόνια των γενεθλίων μας και η συζήτηση αυτή είναι κρίσιμη, θεμελιώδου σημασία. Το έτος της πολιτιστικής κληρονομιάς με ένα πλήρες πρόγραμμα, πολλές εκδηλώσεις, που μάλλον θα κορυφωθούν με την ανακοίνωση της πρωτεύουσας μας ε, Βίλνιους, ε, έναν από τους πιο σημαντικούς προορισμούς ε, για τον πολιτισμό, όπως και το Κάουνας, που έχει θαυμάσια επίσης πολιτιστική παρουσία και έχει ανακοινωθεί ως πολιτιστική πρωτεύουσα για το 2022. Σας καλώ να κλείσετε ήδη για την επίσκεψή σας το 2022. Τέλος πάντων, πέρα από τα αστεία, είχαμε εκδηλώσεις υπό τον τίτλο «Μοντερνισμός για το μέλλον». Και όλα αυτά δεν ήταν ε, στα πλαίσια ενός προγράμματος εθνικιστικής ενότητας, ήταν εστιαζόντουσαν στην τοπική ταυτότητα, στην τοπική παράδοση με τον πιο ουσιαστικό τρόπο. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή. Ευχαριστώ όλους. Α, ξεπέρασα το λεπτό. Ε, βλέπετε τι γίνεται στις Ολομέλειες. Εμείς το πολύ ένα λεπτό έχουμε συνήθως. Είναι τι να κάνουμε, το πεπρωμένο μας εδώ στο Κοινοβούλιο. Λοιπόν, Μαρή Λουίς Οντόνελ από την Ιρλανδία. Για την εκπαίδευση θα μιλήσω. Εντάξει, θα τα κάνουμε αργότερα λοιπόν, θα παρέμβετε μετά. Πάμε να ακούσουμε τον Δημήτριο Σεβαστάκη από την Ελλάδα. Έκανε χθε δύο παρεμβάσεις ε, για το θέμα αποκατάσταση, συντήρηση. Νομίζω όμως ότι μας πάει η συζήτηση και αυτή η καταπληκτική συζήτηση που έχει ε, διεξαχθεί αυτές τις ε, δύο μέρες ε, σε ερωτήματα πολύ πιο ορυκτά και δομικά. Υπάρχει μια κρίση, ιδεολογική κρίση, στον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε την ιστορία και παραλαμβάνουμε το πολιτιστικό απόθεμα. Αυτό το εισήγαγε η νεωτερικότητα. Απ' την άλλη πλευρά η νεωτερικότητα μας άνοιξε τα εργαλεία με τα οποία μπορούμε να κατανοήσουμε βαθύτερα τον πολιτισμό και την ταυτότητα. Και αυτό μας πάει στο εξή. Επειδή υπάρχει μια μεγάλη πολιτιστική αγωνία με τις διασταυρώσεις σήμερα, με τις μετακινήσεις πληθυσμών, αγωνία ταυτότητας, αγωνία ε, αυτοπροσδιορισμού, ακριβώς γι' αυτό το λόγο η πολιτιστική ανάγνωση, το κληροδότημα, το παρελθόν, ο χρόνος μπορεί να γίνει εργαλείο συνοχής από εργαλείο διαίρεσης ε, στο οποίο εξωθούν διάφορες ομάδες και διεθνή λόμπις. Είναι πολύ σημαντικό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, κάνει αυτή τη συζήτηση, θα μου επιτρέψετε να πω, πολυτελείας, ιστορικής, ε, πολιτιστικής πολυτελείας σκέφτεται πάνω σε μεγάλα ανθρωπιστικά επίδικα, όπως είναι ο πολιτισμός, σκέφτεται πώς θα τα εντάξει μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα και σκέφτεται με ποιο τρόπο θα μπορέσει να συμφιλιώσει όχι μόνο τους λαούς με το δικό τους χρόνο, τον ιστορικό χρόνο και το απόθεμα, αλλά πώς θα μπορέσει αυτή η συμφιλίωση να σημάνει μια ευρύτερη συνέβρεση, μια ευρύτερη διασύνδεση. Νομίζω στην δύσκολη και αγωνιώδη πορεία μας για την ενοποίηση της κοινή μας πατρίδας, νομίζω ότι αυτά τα ερωτήματα και αυτές οι συζητήσεις είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Βέσλα Μπερίκοβιτς από το Κροατικό Κοινοβούλιο. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να χαιρετήσω την Επιτροπή Πολιτιστικών Θεμάτων του Κροατικού Κοινοβουλίου, της οποίας είμαι μέλος, και ήθελα να σας παρουσιάσω κάποιες από τις ε, δραστηριότητες ε, και διατάξεις στις οποίες προχωρήσαμε στα πλαίσια της πρωτοβουλίας για την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Πράγματι δεν έχουμε καθόλου χρόνο, αλλά ε, ήθελα να πω ότι έχουμε έναν φορέα, έναν οργανισμό που ασχολείται με την διοργάνωση όλων των εκδηλώσεων στα πλαίσια του πολιτιστικού έτους της ευρωπαϊκής δηλαδή κληρονομιάς, αυτός ο φορέας ε, υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και διοργανώνει περί τις 60, διοργάνωσε περί τις 60 εκδηλώσεις ε, με ευρεία συμμετοχή χιλιάδων ε, πολιτών, εργαστήρια, εκθέσεις Ε, αναλόγως προς τις ε, θεματικές ε, που είχαν προβλεφθεί από το ευρωπαϊκό έτος. Στις δραστηριότητες αυτές συμμετείχαν και τα σχολεία, ενσωματώνοντας στα σχολικά τους προγράμματα εκδηλώσεις και θεματικές. Και είναι πολύ σημαντικό πράγματι οι νέοι και τα παιδιά να διδάσκονται και να αντιλαμβάνονται τη σημασία της πολιτιστικής ε, κληρονομιάς που είναι μέρος ε, της ε, ταυτότητας της ευρωπαϊκής μας. Ελπίζω στο δεύτερο πάνελ να έχω λίγο περισσότερο χρόνο, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα στην κυρία Μπίλτ από τη δική μας την ομάδα. Ένα λεπτό και εσείς. Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτικής Κληρονομιάς ε, έφερε στο προσκήνιο την διατήρηση των ιστορικών κτηρίων. Ε, στην Γαλλία έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό τέτοιων κτηρίων αλλά και τοποθεσιών ε, παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ε, το πρόβλημα δεν είναι τόσο οικονομικό γιατί έχουμε χορηγούς. Ε, υπάρχουν όμως ε, προβλήματα σε κάστρα και παλιά κτίρια εκτός των αστικών κέντρων στην περιφέρεια της Γαλλίας. Για παράδειγμα, στη Γιρόντ, που ένα κάστρο που καταστράφηκε κατά λάθο από έναν ξένο ε, από μια εταιρεία που δούλευε για ένα ξένο καινούριο ιδιοκτήτη. Δεν θα πρέπει να έχουμε λοιπόν καινούριε κατευθυντήρε γραμμέ προ αυτή την κατεύθυνση τη διατήρηση των παλαιών κτηρίων. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε τώρα στην κυρία Πόποβιτς από το Βουλή του Μαυροβουνίου. Ο κύριος Πόποβιτς. Thank you. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ ε, για τη δυνατότητα αυτή να τοποθετηθώ και εγώ συνήθως στο κοινοβούλιο μας είναι η τα μέλη τοποθετούνται για 20 λεπτό είναι πολύ δύσκολο να τους σταματήσει κανείς εδώ έχω πίεση εμείς ε, στο Μαυροβούνιο ήμασταν πάντοτε στην ε, μεθόριο μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών αυτό το έτος ε, της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς είναι πολύ σημαντικό για εμάς γιατί δείχνει τον συσχετισμό, τη διασύνδεση μεταξύ των πολιτισμών των δυτικών και των ανατολικών. Έχουμε διαφορετικές παραδόσεις. Ναι, στο, στο Μαυροβούνιο έχουμε τέσσερις ε, ε θρησκείες, λέει ο μιλητής. Και ίχνη, ε, επιρροές ε, ε, αυστροουγγρικές, ρωσικές και τα λοιπά. Το πλούτος του πολιτισμού μας και της παράδοσής μας σε αυτό ακριβώς έγκυται και από αυτό αντλεί. Νομίζω ότι η ενότητα εντός της διαφορετικότητας που είναι και το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί και πρέπει να εφαρμόζεται και για τη χώρα μας, το Μαρβοβούνιο. Ε, γιατί όλοι μοιραζόμαστε αυτήν την ευρωπαϊκή ταυτότητα και παράδοση χωρίς την οποία δεν θα ήμασταν εμείς το Μαυροβούνιο αυτό που είμαστε σήμερα. Είναι απτά παραδείγματα της σημασίας αυτής της παράδοσης, αυτής της πορείας που μας πέρασαν οι γενναίες του παρελθόντος και φιλοδοξούμε να τις περάσουμε στις επόμενες γενναίες. Σας. Ευχαριστώ. Εμείς ούτε οι πρόεδροι των πολιτικών ομάδων στην Ολομέλεια δεν έχουν 20 λεπτά στη διάθεσή τους για να μιλήσουν. Ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας και πάμε στον επόμενο. Habe ich gerade nicht. Dann kommen wir zu Mrs. Cortez. Η κυρία Κορτέζη από το Κόσο, από το Κοσυφοπέδιο. Good morning to everybody, dear ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να σας παρουσιάσω με λίγα λόγια την κατάσταση της πολιτικής κληρονομιάς και την εκπαίδευση στη δημοκρατία του Κωσυφοπεδίου. Η πολιστική ποικιλομορφία στο Κωσυφοπέδιο είναι ε, κάτι για το οποίο είμαστε περήφανοι. Ήδη το Σύνταγμά μας την προστατεύει. Η πολιτική κληρονομιά προστατεύεται και διατηρείται και μέσω του νόμου πολιτικής κληρονομιάς του Κωσυφοπεδίου και μέσω της δημιουργίας ειδικών προστατευόμενων ζωνών. Παρ' όλα αυτά αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, όπως δεν έχουμε ακόμα επαρκή ε, ένταξη της πολιτικής οικονομία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σε ό,τι αφορά τη λογοτεχνία, μελέτες έχουν δημοσιευθεί για την Συγγνώμη, σε ό,τι αφορά τα επιστημονικά συγγράμματα έχουν δημοσιευθεί πολλές μελέτες για την σημασία της ε, πολιτιστικής μας Είμαστε μια χώρα η οποία βγήκαμε από, μια, από ένα πικιοκρατικό καθεστώς της Σερβίας. Από την άλλη μεριά η πολιτιστική μας κληρονομιά είναι πλούσια και φτάνει στους αρχαίους χρόνους, από τους αρχαίους χρόνους μέχρι τον ε, πόλεμο της απελευθέρωσης της δεκαετίας του 90. Η δημοκρατία του Παιδίου... περιλαμβάνει διάφορες εθνοτικές μειονότητες, όμως οι Αλβανοί αντιπροσωπεύουν το 92% του πληθυσμού. Η πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή. Ε, παρόλα αυτά, επιθυμούμε οι, όλες οι εθνικές μειονότητες να έχουν χώρο έτσι ώστε να μπορούν να εκφραστούν. Και η πολιτική κληρονομιά μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο γιατί αποτελεί ένα ολόκληρο μοσαϊκό. Η πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή ξανά. Ζητώ συγγνώμη, ήμουν αυστηρή με όλους προηγούμενους, πρέπει να σας διακόψω. Μία φράση ακόμα, όχι, όχι, λυπάμαι πάρα πολύ, δεν μπορώ να σας επιτρέψω. Πρέπει να είμαι δίκαιη σε όλους. Σας έδωσα πάνω από δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην επόμενη τελευταία ομιλήτρια. Σνιζάνα Πάουνοβιτς από το Σερβικό Κοινοβούλιο. Πού είναι? Zahvaljujem se i na minutu i želim da sve uvažene kolege... Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για το γεγονός ότι η πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνας στη Βόρεια Σερβία θα είναι πολιτιστική πρωτεύουσα το 2020, η Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, πολιτιστική πρωτεύουσα το 2020. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Ε, θα φιλοξενήσουμε το θεσμό αυτό στη Σερβία. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Ο συνάδελφός μου αναφέρθηκε σε τραυματικά γεγονότα της ιστορίας μας, σε προβλήματα. Είμαι σίγουρη ότι η Ευρώπη θα μας δώσει απάντηση, έτσι ώστε η πολιτική κληρονομιά της Σερβίας, ακόμα και στη νότια, στο νότιο τμήμα της χώρας, να προστατεύεται. Είμαστε υποχρεωμένοι τώρα να ακούμε εδώ πέρα σχόλια και ιστορίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Τα στοιχεία της UNESCO είναι σαφή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κλείνουμε με όλους αυτούς τους ε, παρεμβαίνοντες ε, το πρώτο πάνελ. Έχουμε άλλα δύο. Στο δεύτερο λοιπόν θεματικό πάνελ θα δούμε τα θέματα της ε, διατήρησης, συντήρησης και αποκατάστασης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ξέρουμε ότι σε όλα τα κρατημέλη είναι μεγάλη πρόκληση αυτό, γιατί πάντα κοστίζει πολύ η αποκατάσταση. Οπότε να ε, δώσω το λόγο στον πρόεδρο του χτεσινού πάνελ για να μας κάνει μια σύντομη περίληψη της χτεσινής συζήτησης. Ο κύριος, ο συνάδελφος Διάκονο έχει το λόγο. Σας ακούμε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, ε επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι στο δυνατόν πιο σύντομος θέλω να πλουστεύσω τα πράγματα, οπότε θα πω ότι έγινε πραγματικά μια εξαιρετική συζήτηση εχθές. Οι ομιλητές παρουσίαζαν πολλές θετικές προκλήσεις και θέλω να επικεντρωθώ σε αυτά που είπαν κυρίως οι προσκεκλημένοι μας, γιατί νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά σε σχέση με το τι λέμε εμείς. Ε, γιατί αυτοί πραγματικά παρουσιάζουν την πραγματικότητα. Η συζήτηση ξεκίνησε με μια συνολική παρουσίαση από την Γενική Διεύθυνση Πολιτισμού ε, που ε, μας παρουσίασε τους βασικούς στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης παρουσίασε τις βασικές πρωτοβουλίες, ε, επικεντρωνόμενοι βεβαίως και στα θέματα της διάσκεψης, ε, δηλαδή αρμοδιότητα για την πολιτιστική κληρονομιά, επιστήμη για την κληρονομιά και διατήρηση της κληρονομιά. Μετά ακολούθησαν οι διάφοροι ομιλητές και κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου ερωταπαντήσεων τονίστηκαν κάποια σημεία, όπως ας πούμε η καταστροφή των της πολιτικής χρονομιάς από φυσικές καταστροφές, η σημασία των επαγγελμάτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση της ε, πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης, η ανάγκη για αλληλεγγύη και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς το πρόβλημα της ε, ανάπτυξης των αστικών κόμβων, η χρήση των διαρθρωτικών ταμείων σε διάφορα κρατημέλη και πώς αυτή σχετίζεται με την πολιτιστική κληρονομιά, κυρίως για την κατανομή των κονδυλίων ώστε να διατηρηθούν, να συντηρηθούν κτίρια. Επίσης, ε, πρόσβαση σε όλους τους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και η χρήση ε, και η αναγκαιότητα της ε, εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Μετά, κατά τη διάρκεια της δεύτερου, του δεύτερου γύρου ερωταπαντήσεων, ακούσαμε θέματα όπως η σημασία της διατήρησης των, χωρών των περιοχών της υπαίθρου και τον, τον πληθυσμό που ζουν εκεί, οι αρχαιολογικοί χώροι χρειάζονται, χρήζουν ειδική προστασία και πρέπει να δημιουργηθεί ένα δίκτυο μεταξύ αυτών των χώρων ώστε να είναι κανεί περήφανο για την κληρονομιά του. Και κατά τη διάρκεια της τρίτης, του τρίτου γύρου ρωταπαντήσεων ακούσαμε ε, την ε, σημασία της ε, χρήσης των ε, κτηρίων, της επένδυσης στον, τουρισμό, συγγνώμη, της ε, αύξησης ευαισθητοποίησης, της εκμάθησης ε, μιας τέχνης που άπτεται του τομέα της πολιτικής χειρονομιάς και βεβαίως πώ όλα αυτά μπορούν να ενταχθούν στις, ε, στα θεματολόγια των κρατών μελών. Ήταν πραγματικά ε, καρποφόρα η συνάντηση αυτή. Όλοι πήραν μέρο, μα ανέφεραν πολύ σημαντικά θέματα, οπότε μπορούμε να προσλέπουμε σε πολύ σημαντικέ εξελίξει. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για την σύντομη και πλήρη και περιεκτική παρέμβασή σας και ευχαριστώ που αναλάβατε την Προεδρία του πάνελ αυτού. Πάμε τώρα στη Σούζαν Κορ. Είναι η πρόεδρος της ΕΚΟ, της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας Οργανώσεων Συντήρησης και Αποκατάστασης. Σούζαν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων συνάδελφοι, σε αυτό το ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς η Ένωση των Οργανώσεων Συντηρητών ε, Μνημείων Τέχνης έχει την τιμή σήμερα ε, να κάνει αυτή την τοποθέτηση στην χρονιά που γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι χρήσιμο να θυμόμαστε τα χρόνια εκείνα και το πώς ε, μας οδηγούν εδώ ε, τι ρόλο διαδραματίζουν στην κοινή μας παράδοση, ε, στην ιστορική μας μνήμη, στα ιστορικά μας αρχεία. Πώς δηλαδή διαμορφώνουμε την ιστορική αλήθεια. Η διαβίβαση λοιπόν ένας, ενός αυθεντικού ε, κληροδοτήματος είναι μια έννοια κλειδί στην καλύτερη κατανόηση της συντήρησης και της αποκατάστασης των ε, μνημείων της ιστορικής παράδοσης. Αυτή η παράδοση είναι μοναδική και αναντικατάστατη και αυτό είναι μια ευρωπαϊκή αξία από μόνο του. Δεν είναι ο σκοπός ε, της συντήρησης των μνημείων να δημιουργήσει νέα στοιχεία, αλλά να χρησιμοποιήσουμε, να μας επιτρέψει δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία της ευρωπαϊκής μας πολιτιστικής κληρονομιάς ως αρχεία ως μνημεία του ιστορικού παρελθόντος. Πρέπει κανείς να εκτιμά λοιπόν διαρκώς ε, την φθορά τους και τον τρόπο της αποκατάστασής τους και διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την ανταπόκρισή μας. Ποια είναι τα επίπεδα της παρέμβασης, πόσο μακριά μπορεί να πάει μια αποκατάσταση ή μια συντήρηση ώστε να παραμείνει τέτοια και να μην είναι επιθετική παρέμβαση σε ένα μνημείο. Και ποια είναι τα στοιχεία της φθοράς και της απώλειας. Πώς τηρούμε στοιχεία, πώς μαθαίνουμε περισσότερα στοιχεία για το παρελθόν. Όλα αυτά είναι τμήμα ενός διαλόγου με τις κοινότητες και με τους υπόλοιπους επαγγελματίες έχουμε εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης ώστε να παρεμβαίνουμε και να σώζουμε, να διατηρούμε αυτήν την, αυτό το κληροδότημα. Ε, αυτά καθοδηγούν τους συντηρητές ε, ε, μνημείων και έργων τέχνης μέσω έρευνας και είναι όλα αυτά στοιχεία δημοσίου ενδιαφέροντος. Εμείς ως Ένωση επιμένουμε ότι ένα συντηρητής μνημείων και ε, έργων τέχνης θα πρέπει να ε, ε, λαμβάνει ένα πτυχίο επίπεδου μάστερ. Η ΕΚΟ είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο εθνικών ενώσεων και φορέων που θέτει βέλτιστες πρακτικές προσπαθώντας να εξασφαλίσει την ύψιστη δυνατή ποιότητα για την εκπαίδευση των συντηρητών και την διαμόρφωση ε, κατευθυντηρίων γραμμών για τις δεξιότητες των ε, τεχνητών αυτών. Αυτά θα πρέπει να διέπονται από νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. Πρόσφατα είχαμε και την πρώτη ημέρα της Ευρωπαϊκής Συντήρησης Μνημείων τον Οκτώβριο με εργαστήρια και εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη ώστε να υπογραμμίσουμε την αξία και την σημασία της δουλειάς αυτής που γίνεται η Ευρώπη είναι ένα παλίψιστο υλικών στοιχείων με, διάφορα, με διάφορες παραδόσεις. Όλα αυτά συνθέτουν το πλαίσιο των ευρωπαϊκών αξιών και αυτό αποτυπώνεται και στον υβριδικό τίτλο Conservator Restorer, συντηρητής αποκαταστάτης. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα στοιχεία μνήμης και παράδοσης θα διαβιβάζονται ανώθευτα στο μέλλον. Ο τομέας ε, του πολιτισμού με τις διάφορες εκδηλώσεις του ε, αποτυπώνεται ελιπέστατα στις διάφορες οικονομικές ερευνές που έχουμε γιατί είναι πολύ σημαντικός για τη διαβίβαση γνώσεων και δεξιοτήτων για τα προγράμματα εκπαίδευσης. Ζητούμε η Επιτροπή Πολιτισμικών Θεμάτων να υποστηρίξει τις προσπάθειες αυτές μέσω των πορισμάτων από την ε, ομάδα ανοιχτής μεθόδου συντονισμού σε αυτό το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στα πλαίσια του θεματολογίου για τον πολιτισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Κυριάκο Χατζηγιάννη, μέλος του Κυπριακού Κοινοβουλίου και πρόεδρο της Επιτροπής ε, Πολιτισμού. Σας ακούμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, είναι με ιδιαίτερη χαρά που μπορώ να προσφωνώ αυτή τη διάσκεψη για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα. Καταρχήν, θα ήθελα να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εξαιρετική του αυτή πρωτοβουλία να ανακηρύξει το 2018 σε ένα ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς. πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης αποτελεί το, το πολύτιμο κοινό πόρο. Περιλαμβάνει την κοινή ιστορία μας και τις αξίες μας, τα οποία αποτελούν τον πυρήνα του σχεδίου της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ένα πλήγμα ενάντια στην ταυτότητα αλλά και την ιστορία των πολιτών μα και τη παγκόσμια κληρονομιά τη ανθρωπότητα. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι ευάλωτη, ιδιαίτερα σε περιόδου ένοπλων συγκρούσεων. Η αξία και η σπανιότητα αρκετών πολιτιστικών αντικειμένων τα εκθέτει στον κίνδυνο παράνομη μετακίνηση από αρχαιολογικού χώρου, κλοπή από μουσεία, παράνομη εμπορία αλλά και πώληση. Είναι προφανέ ότι σε περιοχές με παρατεταμένες συγκρούσεις, η πολιτιστική κληρονομιά θυματοποιείται, καθώς η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών επιδεινώνεται, πόσο μάλλον η φυσική καταστροφή των θησαυρών και των ιδίων των τόπων μας, γεγονός το οποίο αποτελεί μη ανατρέψιμο γεγονός. Η διεθνής κοινότητα έχει κλονιστεί πρόσφατα από τις συγκλονιστικές εικόνες της βίαιης καταστροφής πολιτιστικών και ιστορικών χώρων κατά την παράνομη εμπορία τους από το Ισλαμικό κράτος στη Συρία και το Ιράκ. Οι συγκεκριμένοι χώροι αποτελούν μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ιστορικοί χώροι έχουν υποστεί ζημιά συνεπία βομβιστικών επιθέσεων αλλά και βανδαλισμών. Το παράνομο εμπόριο λαϊλατημένων πολιτιστικών αγαθών από τη Συρία και το Ιράκ ευδοκιμεί. Η διεθνής κοινότητα έχει υιοθετήσει σχετικά ψηφίσματα που καταδικάζουν αυτέ τι ενέργειε, χαρακτηρίζοντά τι ω έγκλημα πολέμου. Αυτέ οι καταστροφέ αποτελούν ανεπανόρθωτε απώλειε για τι μελλοντικέ γενιέ τη ανθρωπότητα στο σύνολό τη. Είναι καθήκον μα λοιπόν να διαφυλάξουμε ό,τι μπορεί ακόμη να διασωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η έκταση και η βαρβαρότητα τη καταστροφή τη πολιτιστική κληρονομιά στη Συρία και το Ιράκ απαιτούν προβληματισμό σχετικά με τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την αποτελεσματική προστασία τέτοιων θησαυρών. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω τη Σύμβαση για τα αδικήματα που σχετίζονται με πολιτιστικά αγαθά που υιοθετήθηκε το 2017 στο πλαίσιο τη Κυπριακή Προεδρία τη Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Η Σύμβαση αποτελεί ορόσημο στην ποινικοποίηση τη παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών. Δράττω με τη ευκαιρία να ενθαρρύνω όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να ασκήσουν ανάλογη πίεση στις εθνικές κυβερνήσεις τους για επικύρωση αυτής της σύμβασης προκειμένου να ενδυναμωθούν οι προσπάθειές μας προς αυτή την κατεύθυνση. Η Κύπρος προσδίδει μεγάλη σημασία στο ζήτημα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, αναγνωρίζοντας ότι οι αρχαιότητες αλλά και άλλα ιστορικά και πολιτιστικά αγαθά αποτελούν το συνδετικό κρίκο των λαών με το κοινό τους παρελθόν, καθώς ενισχύει και το κοινό αίσθημα το πού ανήκει κάποιο. Συνεπία τη τουρκική εισβολή του 1974, η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του καχτεκόμενου τμήματο του νησιού έχει υποστεί σημαντικέ ζημιέ και ορισμένα μνημεία κινδυνεύουν με πλήρη εμφανισμό. Εκατοντάδε εκκλησία, μοναστήρια, άλλα θρησκευτικά μνημεία και νεκροταφεία έχουν λαιλατηθεί, βεβηλωθεί και κατεδαφιστεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 44 ετών. Αρχαιολογικά μουσεία έχουν λαιλατηθεί και αρχαιολογικές συλλογέ εκτίθενται στις διεθνεί αγορές. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών, θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παροχή σημαντικής οικονομικής στήριξης στις εργασίες της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά. Από το 2012, χάρη στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, UNDP, η Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά έχει συντηρήσει, υποστηρίξει δομικά, αναστηλώσει ή αποκαταστήσει 31 έργα πολιτιστικής κληρονομιάς σε ολόκληρο το νησί, περιλαμβανομένων Ορθοδόξων, Μαρονίτικων και Αρμένικων εκκλησιών, τζαμιών, μιναρέδων, οχυρώσεων, χαμάμ, υδραγωγείων και νερόμυλων. Το έργο της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα αγαστής συνεργασίας μεταξύ των Κυπρίων, Έλληνο-Κυπρίων και Τουρκοκυπρίων, με κοινό σκοπό και αμοιβαίο σεβασμό για τη διαφύλαξη τη κοινή του κληρονομιά. Ωστόσο, με λύπη μου, σα πληροφορώ ότι σύμφωνα με πρόσφατε αποκαλύψει στον τουρκοκυπριακό τύπο, μεγάλο αριθμό ελληνοορθόδοξων εικόνων και άλλων θρησκευτικών αντικειμένων παρέμειναν παγιδευμένα στο κάστρο τη Κερίνια από την τουρκική εισβολή του 1974. Υπάρχουν σοβαρέ ανησυχίε σχετικά με τη σωστή του φύλαξη, τη συντήρηση και την προστασία του καθώ και λόγω τη υγρασία που επικρατεί στην τοποθεσία λόγω τη εγκύτητά τη με τη θάλασσα. Κάνω έκκληση στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να επιδείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη του, ασκώντα την απαραίτητη πίεση στην Τουρκία για την επιστροφή αυτών των πολιτιστικών θησαυρό στον νόμιμο ιδιοκτήτη του που είναι η Ορθόδοξη, Ελληνική Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία τη Κύπρου. Καταλήγοντα, θα ήθελα να τολίσω ότι είναι ύψη τη σημασία η κινητοποίηση και επένδυση περισσότερων κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως μέσω του προγράμματος Ορίζοντας 2020 για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς για την προστασία και διατήρηση της κληρονομιάς όλης της ανθρωπότητας για τις μελλοντικές γενιές. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ich möchte wirklich noch mal alle θα ήθελα να ζητήσω παρακαλώ από όλους να τηρείτε τον όρο αγόρευσης, γιατί αλλιώς θα φύγουμε τελείως από το πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε σε άλλον έναν πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτισμού της Γερουσίας της Ρουμανίας. Ράντου Κόσμιν Πρέντα. Σας ακούμε. vreau să vă spun câteva Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σα πω δύο πράγματα για την ρουμανική πολιτιστική κληρονομιά. Στα πλαίσια και της, ε, του εορτασμού των 100 ετών. Ε, καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για την ε, διεξαγωγή αυτής της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής γιατί μας δίνει την δυνατότητα να συζητήσουμε ένα από τα πολύ σημαντικά θέματα της ευρωπαϊκή ταυτότητα στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η Ευρώπη έχει μια ιστορία πολιτισμού και ο πολιτισμό είναι αυτό που ενώνει τα κράτη μα ε, πάνω σε κοινέ ε, αξίε που μπορούν να συγχωνεύσουν τις ε, διαφορετικές ιδιαιτερότητες των κρατών μελών. Πρέπει λοιπόν να συνεχιστεί ο διάλογος μεταξύ των κρατών μελών αλλά και μεταξύ των κρατών μελών και, της, και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση αυτό, ε, καλωσορίζουμε βεβαίως τις δραστηριότητες που οργανώνονται στα πλαίσια της ε, ε, πολιτικής κληρονομιάς. Εμείς διοργανώνουμε τέτοιες δραστηριότητες και τα μνημεία που υπάρχουν στην Ρουμανία είναι πραγματικά πολύ σημαντικά είναι σημαντικά σύμβολα αξιοπρέπειας της ε, Ρουμανίας. Ε, στα πλαίσια του 2018 Έχουμε επίσης δύο πτυχές που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Καταρχάς ότι το 2018 είναι το έτος πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και ότι έχουμε την, ε, τα 100 χρόνια εορτασμού της ενοποίησης της Ρουμανίας. η πολιτιστική κληρονομιά βεβαίως είναι σημαντικό κομμάτι της ιστορίας μας, ε, της ε, ιστορικής μας ταυτότητας, της σύγχρονης ταυτότητας της Ρουμανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια λοιπόν του εορτασμού ε, έχουμε διάφορες δραστηριότητε που ασχολούνται με την συμμετοχή όλης της κοινωνίας της Ρουμανίας, του τοπικού επίπεδου, της περιφέρειας, των τοπικών κοινοτήτων. Ένα κομμάτι της... Ε, ένα κομμάτι των εορτασμών βεβαίω ε, αφιερώνεται και στα 100 χρόνια από την ενοποίηση. Φυσικά πρέπει να έχουμε στα χέρια μα ε, στρατηγικέ και εργαλεία για να υπάρχει καλύτερη συμμετοχική δημοκρατία, συμμετοχή ερευνητών στι πολιτικέ και όσων ασχολούνται με το θέμα τη πολιτική κληρονομιά σε ό,τι αφορά τώρα την, την κληρονομιά από τις εθνικές μειονότητες και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ε, του πολιτισμικού, πολυπολιτισμικού προφίλ που έχει η Ρουμανία και εφαρμόζοντας τις ε, πρωτοβουλίες αυτές σύμφωνα και με την, νομικέ ε, τις νομικές πράξεις της Ένωσης μπορούμε να προστατεύσουμε την ταυτότητα με, που βασίζεται στην πολιτιστική ποικιλομορφία. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι και ηλική κληρονομιά και πνευματική και αποτελεί την πηγή που μπορεί να μας βοηθήσει στο μέλλον. Γι' αυτό η κληρονομιά πρέπει να μεταλαμπαδευτεί στις επόμενες γενναίες για να μπορέσουν να την αναπτύξουν. Πρέπει βεβαίως να έχουμε υπόψη ε, τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν και οι οποίες πρέπει να προστατευθούν μέσω καινοτόμων προσεγγίσεων, ανταλλαγής εμπειριών, ιδεών και καλών πρακτικών το διοικητικό πλαίσιο με βάση το διάλογο και θα πρέπει να βασιστεί στο διάλογο και την ευέλικτη νομοθεσία. Στην Ρουμανία ασχολούνται διάφορες υπηρεσίες ε, με την, ε, με την κατανομή των κονδυλίων που δίνονται για την αποκατάσταση των ιστορικών μνημείων από το ε, κράτος. Το, το σχετικό Ινστιτούτο έχει διοργανώσει διάφορες ε, συζητήσεις, πάνελ, για να γίνει μια μελέτη της κατάστασης των πολιτιστικών μνημείων και να καταγράψει διάφορα έργα που θα μπορούσαν να αποκατασταθούν. Πρόσφατα στην ε, νομοθεσία μας υιοθετήσαμε τα σχετικά στοιχεία ώστε να υπάρχουν ε, οι οικονομικοί πόροι για να μπορούμε να μεταφέρουμε και την οδηγία του 2014-2016 για την αποκατάσταση των ε, ε, πολιτιστικών αγαθών που παράνομα αφαιρούνται από την επικράτεια των κρατών μελών. Επίσης, ε, τροποποιήσαμε την εθνική μας νομοθεσία έχοντας ένα εθνικό κεντρικό μητρό κινητών αγαθών που εμπίπτουν σε ειδικά προγράμματα. Η Ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης επίσης έδωσε τη δέουσα προσοχή στα θέματα κληρονομιάς και αξιολόγησης, εφαρμόζοντας ε, βεβαίως ε, το Ευρωπαϊκό έτο πολιτιστική Κληρονομιάς. Η κληρονομιά θα ε, αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της πολιτικής μας και θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι πρέπει να δούμε και, τα, την απτή και την άλλη κληρονομιά μας. Ευχαριστώ. Vielen herzlichen Dank auch Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση αυτή. Πάμε τώρα στην Ιρένα Στεφόφσκα. Είναι πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Εκπαίδευσης στο Κοινοβούλιο της ΦΥΡΟΜ. Πού είστε, σας ακούμε. Ladies and Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, ε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα να μιλώ εκπροσωπώντας ε, την δημοκρατία της Μακεδονίας, της Βόρειας Μακεδονίας. σχετικά με την περίπλοκη και πολυσύνθετη παράδοση την ιστορική. Αυτή αποτυπώνεται σε διάφορα αρχιτεκτονικά μνημεία, μνημεία των καλών τεχνών, βιβλία, συγγράμματα. Όλα αυτά μας προσφέρουν πολλαπλές δυνατότητες ε, για την ε, συμπερίληψή τους στην καθημερινή μας ζωή και την καλύτερη κατανόησή τους. Και σε μια συζήτηση του τι επιθυμούμε να κάνουμε σχετικά με την παράδοση αυτή. Και τι είναι η παράδοση αυτή για τη χώρα. Ένα τουριστικό προϊόν που θέλουμε να εκμεταλλευτούμε ή είναι ένα απόσπαστο κομμάτι ε, μιας, ε, ενός τρόπου ζωής ε, πολιτισμένου, αστικού. Είναι μια αναγκαιότητα, είναι ένα αγαθό. Χρειάζεται λοιπόν ένα πλαίσιο παιδείας ένα πλαίσιο διατήρησης αυτού του περιβάλλοντος προκειμένου να προστατεύσουμε, να διαχειριστούμε και να προσφέρουμε μεγαλύτερη επιφάνεια σε αυτά τα στοιχεία. Το πολιτιστικό πλαίσιο στην ε, δημοκρατία της ε, Μακεδονίας ε, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των αγαθών αυτών ούτε σε παγκόσμιες πρακτικές. Εμείς προσπαθούμε να δουλέψουμε επί ενός προτύπου προτεραιοποίησης των στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς και η τοποθέτησή τους σε ένα ευρωπαϊκό ευρύτερο πλαίσιο. Το πιο σημαντικό ζήτημα στην δική μας περίπτωση είναι πώς ε, ταυτόχρονα θα επιτύχουμε την προστασία τους, την αποτελεσματικότητα των φορέων που θα είναι υπεύθυνοι για την προστασία αυτά και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τη σημασία του κληροτήματος του πολιτιστικού. Το πρότυπο αυτό επί του οποίου εργαζόμαστε συνδέεται με την Εθνική Στρατηγική Πολιτιστικής Ανάπτυξης για την περίοδο 18 έως 22. Λόγω της υψηλής αποτελεσματικότητας των σχετικών φορέων, η Επιτροπή Πολιτιστικών Θεμάτων παρενέβη με εννέα τροπολογίες στο τμήμα της στρατηγικής που ακριβώς αναφερόταν στην προστασία των ε, ε, μνημείων της πολιτιστικής ε, κληρονομιάς. Η Επιτροπή της οποίας προεδρεύω διοργάνωσε μια ακροματική διαδικασία σχετικά με τις διατάξεις των τοπικών κυβερνήσεων της περιοχής Όχριτ που είναι και στην, ε, έχει εγγραφεί ως παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά από την UNESCO. Οι τοπικές λοιπόν ε, οι τοπικοί φορείς και οι τοπικές κυβερνήσεις θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το πρότυπο. Η Διεύθυνση για την Προστασία των Αγαθών Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι ανεξάρτητος φορέας που είναι υπεύθυνο για την ε, επιβολή, την υλοποίηση του κανονισμού σχετικά με τα μουσεία και, τα, και τους χώρους πολιτιστικής ε, κληρονομιάς. Είμαστε εν μέσω μιας διαδικασίας αποκέντρωσης του συστήματος προστασίας και διαφοροποιούμε μεταξύ τριών συνιστοσών οι οποίες θα πρέπει να αποτυπωθούν στο όλο θεσμικό πλαίσιο που είναι τα μουσεία, τα, η προστασία και η έρευνα και βεβαίως η παιδεία. Η εκπαίδευση. Αυτή είναι, αυτές οι συνιστώσεις είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους αλλά και διασυνδεδεμένες και είναι ανοιχτές προς τις παγκόσμιες πρακτικές. Το Υπουργείο Πολιτισμού είναι ο φορέας που ενώνει αυτές τις συνιστώσεις αυτή τη στιγμή, αλλά θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και την δημιουργία ενός ε, ανεξάρτητου, ενός νέου θεσμού που θα εστιάζεται ε, στα στοιχεία του πολιτισμού το οποίο θα επιτρέψει μια καλύτερη επαγγελματική αρεστία και καθοδήγηση στην έρευνα και των λοιπόν δραστηριοτήτων που συνιστούν την προστασία των, της πολιτιστικής κληρονομιάς. δεδομένη της υποψηφιότητα που έχει η χώρα, όλα αυτά θα πρέπει να προχωρούν παράλληλα με τα κριτήρια της Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τη συμμόρφωση προ αυτά, δηλαδή ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία τη πολιτική κληρονομιά, η βελτίωση της αριστείας ε, και η συμμετοχή των πολιτών, του κοινού. Είναι σημαντικό επίσης να ανταλλάσσουμε εμπειρίες με άλλες χώρες και, και τέλος μην ξεχνούμε ότι η παράδοση σχετίζεται με τους ανθρώπους, με τους πολίτες Αυτό που κάνουμε ως ε, πολιτικοί, επαγγελματίες, ε, τεχνικοί Θα πρέπει να το κάνουμε για τους πολίτες ώστε αυτοί να συμμετέχουν στο, στην ε, απόλαυση αυτής της παράδοσης και αυτών των μνημείων. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Εγώ ε, ευχαριστώ. Πάμε στον τελευταίο παρεμβαίνοντα. Και εδώ πάλι έχουμε έναν πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτισμού της Γερουσίας της Πολωνίας. Ο κύριος Γέρζη Φεντερόβιτς. Πού είστε? Εκεί είστε. Έχετε το λόγο. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Postaram się zmieścić, bo ja... Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω από στήθους, δεν έχω κάτι γραμμένο, έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις από αυτά που ήθελα να πω. Συμφωνώ με όλα όσα είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Ε, καταρχήν, η κουλτούρα, ο πολιτισμός αντικατοπτρίζει την ταυτότητα. Και είναι πολύ καλό που λαμβάνει η χώρα τώρα αυτή η συνάντηση στην ε, Πολωνία. Ε, καταφέραμε να πετύχουμε την ανεξαρτησία μας ε, πρόσφατα σχετικά και χάρη στην κουλτούρα μας, χάρη στους συγγραφείς μας, τους συνθέτες μας, τους ανθρώπους των γραμμάτων. Η κουλτούρα είναι ελευθερία. Και θα ήθελα να εστιάσουμε σε αυτό που είπαμε πριν. Η κουλτούρα δεν θα πρέπει να είναι ένα εργαλείο βίας, δεν θα πρέπει να είναι ένα εργαλείο ξενοφοβίας, ρατσισμού, ή μίσους. Είναι πολύ σημαντικές οι μέρες πολιτικής κληρονομιάς. Πρέπει να επωφεληθούμε από αυτό το θεσμό για να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή κουλτούρα σε όλο τον κόσμο και για να φτάσουμε στην ολοκλήρωση που επιθυμούμε. Πρέπει να ευχαριστήσω όλη την Ευρώπη μετά από πολλά χρόνια κομμουνισμού χάρη στην, στον πολιτισμό καταφέραμε να απελευθερωθούμε. Τότε ήμουν ηθοποιός και σκηνοθέτης, θεατρικός σκηνοθέτης και εργαζόμουν με ανθρώπους που η ελευθερία ήταν πάρα πολύ σημαντική για αυτούς. Τον ε, Αντρέι Βάιντα για παράδειγμα, ο Κισλόφσκι, ε, αυτοί οι σκηνοθέτες που έδειχναν πως η κουλτούρα μπορούσε να μας βγάλει από το κομμουνιστικό σύστημα. Και τελικά το καταφέραμε και ενωθήκαμε με την Ευρώπη. Χάρη στην ε, βοήθειά σας, ε, χάρη στα, τη βοήθεια, την οικονομική και άλλη βοήθεια που ήρθε από την Ευρώπη, καταφέραμε να χτίσουμε για παράδειγμα το κέντρο ελεγγύης του Γκτάνσκ, το μουσείο της ε, μουσικής της, του Μπρέσλαβ, Όλα αυτά σε μεγάλο βαθμό είναι επιτεύγματα χάρη στην οικονομική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι δεν θα πρέπει να, ρωτάμε την, να ζητάμε από την Ευρώπη αυτά που θέλουμε από εκείνη. Πρέπει πρώτα να δούμε εμείς τι μπορούμε να προσφέρουμε στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι κάνουμε πολλά για την Ευρώπη και εμείς. Για παράδειγμα, τα, το φεστιβάλ ε, εβραϊκής κουλτούρας που διοργανώνουμε, ε, το έργο το οποίο ε, δωρήσαμε για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την, τις διασυνοριακές επαιτίους και εκδηλώσεις για, την εβραϊκή, για τον εβραϊκό πολιτισμό με γειτονικέ χώρες. Αυτά είναι παραδείγματα για να καταλάβετε πώς συνεισφέρουμε εμείς ε, στην ε, Ευρώπη. Επίσης, ε, έχουμε πάρα πολύ τεχνογνωσία σε θέματα συντήρησης Έχουμε τεχνικές τις οποίες εμείς ανακαλύψαμε και χρησιμοποιούν πια σε όλο τον κόσμο. Μερικές φορές βέβαια λένε, ότι, ε, λέγεται ότι ο πολιτισμός δεν είναι επαρκώς ε, παρόν, είναι αλήθεια. Μερικές φορές μάλιστα ε, ο πολιτισμός γίνεται και αντικεί, εμπορικό αντικείμενο, εμπορευματοποιείται. Στην ε, Κρακοβία, για παράδειγμα, έχουμε παρόμοια προβλήματα με αυτά τη βενετία λόγω του τουρισμού. Έγινε μια συνάντηση τη ε, UNESCO σε σχέση με την, τον πολιτισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ την UNESCO γι' αυτό. Και εκεί συμμετείχαμε πολλοί από, συμμετείχαν πολλοί από αυτούς που είναι εδώ, ο κ. Γκουτιέρεθ για παράδειγμα, πολύ βουλευτές, ευρωβουλευτές ε, και θα ήθελα να πω και στη συνάλφω από τη Μακεδονία ότι έχουμε συνεργαστεί με τα Σκόπια για την συντήρηση αμφιθεάτρων εκεί πέρα. Έχω ξεπεράσει το χρόνο μου, αλλά έχω άλλη μια έκπληξη, γιατί είμαι, όπως σας είπα, ηθοποιός και υπάρχουν και άλλοι ηθοποιοί εδώ μέσα θα ήθελα να σας προσκαλέσω σε μια εκδήλωση, να πω το εξής. Ε, ένας Πολωνός ποιητής έχει γράψει ένα ποίημα με ομοιοκαταληξία, ε, πέθανε σε, σε, ε, του συγκέντρωσης. Ε, πρέπει να διαβάσει μια φορά κανείς, πρέπει να διαβάσει δυο φορές, πρέπει να διαβάζει για χρόνια και μόνο έτσι θα φτάσει το πουλί να φάει ψίχουλα από την παλάμη του. Που που πετάει μπροστά σου. Πρέπει να γράψεις μια φορά, δυο φορές, πρέπει να γράφεις για χρόνια μέχρι ότου το πουλί αυτό να προσγειωθεί στο χέρι σου και να σε γλιτώσει από τη μοναξιά σου. Να, μέχρι να σε πάρει μακριά πάνω από βουνά και ποταμούς. Πίστεψε Εμπιστέψου τον εαυτό σου, ξεκίνα από την αρχή γιατί έτσι ξεκινάει ο κόσμος. Αυτό ήταν το ποίημα σε ελεύθερη μετάφραση. Ευχαριστούμε πολύ και για αυτή την πολιτιστική ποιητική παρέμβαση. Πάμε τώρα στην, στον κύριο συζήτησης. Πάλι εννέα έχουν ζητήσει το λόγο. Πάλι θα σας περιορίσω στο ένα λεπτό τον καθένα και ξεκινούμε με τον πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτισμού της ε, Ιταλικής Βουλής. Πού είστε? Παρακαλώ, σας ακούμε. Γκάλο. Καλημέρα Πρόεδρε, καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι και προσκεκλημένη είναι μια χρυσή ευκαιρία να μιλούμε για ένα στρατηγική σημασία θέμα για την Ευρώπη που είναι ο πολιτισμός ε, και η παιδεία. Θα μπορούσαμε να είμαστε υπερδύναμοι πολιτιστικοί ως Ευρώπη. Η επένδυση στον τομέα αυτό δεν σημαίνει απλώς ε, την ανάπτυξη της οικονομίας, εφιών, ε, πολιτικών που συμβάλλουν και στην απασχόληση, αλλά πραγματικά είναι ένα νέο πρότυπο οικονομικής δραστηριότητας και ανάπτυξης. Και νομίζω ότι έχουμε και απεγνωσμένα την ανάγκη αυτή του, του μοντέλου, γιατί διερχόμαστε μια ε, υπαρξιακής κρίσεως οικονομικής και άλλης που αντιμετωπίζουμε εδώ και καιρό είναι τα στοιχεία που μας δείχνουν σήμερα ότι υπάρχει ένα, ένα πολιτιστικό μάλλον πρότυπο που με την εμφάνιση των, ε, της κρίσης, της απειλής σε όλους τους υπόλοιπους ε, ε, τομείς, ο πολιτισμός είναι αυτός που εξακολουθεί να παρέχει ευκαιρίες και μιλώντας για ανάπτυξη, για μεγέθυνση, πρέπει να προσπαθήσουμε να προσπεράσουμε τα δεσμά που ε, θέτουμε στα ε, πολιτιστικά ε, θέματα υπό τον προϋπολογισμό γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό διαχείριμα για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Επόμενος, ο Ράιναχαρτ Πίζετς, πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού της ε, Βουλής της Αυστρίας. Σας ακούμε. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτικής Οικονομίας 2018 είναι ένα, ένας τρόπος κατανόησης της ιστορίας. Τι έχει γίνει με βάση τα όσα έχουν μείνει πλέον στις ημέρες μας. Θα ήθελα να μιλήσω για την Αυστρία. Έχουμε ε, ξεκινήσει διάφορα project τα τελευταία χρόνια και θέλω να μιλήσω για διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Αν έρθετε στην, στις 6 και 7 Δεκεμβρίου στη Βιέννη, ε, θα δείτε ότι πραγματικά υπάρχει ένα apartheid πολιτιστικό στην, ε, στη Βιέννη. Θα ήθελα να το διερευνήσετε αυτό, γιατί η δόμηση είναι και κρατικό, ε, κρατική νομοθεσία, αλλά και τοπική αλλά πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλές ε, πρωτοβουλίες στην ε, ε, Βιέννη, αλλά 60% των κυμάτων της Βιέννης υπάρχουν από τον 18 19 αιώνα. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε λοιπόν και να προσέξουμε πολύ περισσότερο την πολιτιστική κληρονομιά και όχι τόσο τους κανόνες δόμησης. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε στον Φέλιξ Μόντες Φως από την Ισπανική Γερουσία. Πού είστε? Σας ακούμε. Καλημέρα σε όλους, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η πολιστική κληρονομιά και η παράδοση είναι ε, θεμέλια για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και από τις δεσμεύσεις που χρησιμοποίησαμε για, την, για την περίοδο 14-18 για την καινοτομία και την οικονομία πρέπει να προσθέσουμε την αλληλεγγύη, την αδαφικότητα και τη γέφυρα μεταξύ των γενεών. Και αναφέρομαι και στην ύπεθρο στους πολίτες που κατοικούν εκτός των αστικών κέντρων. Μιλώ για προσβασιμότητα, μιλώ για την ε, ε, ε, ομαδική συλλογική ευθύνη για την ε, ταυτότητα, για την συμμετοχικότητα. Στην ουσία μιλώ για τους ανθρώπους, για τους πολίτες που πρέπει να προστατεύσουμε τα ήθη, τα έθιμα, την εργασία, την παράδοση, την απτή. Δηλαδή των, κατοίκων όλων των περιφερειών και όλων των περιοχών μας. Και πρέπει να το δούμε αυτό ως πόρο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ. Πάλι από, σε μέλος της Επιτροπής μας εδώ, η Julie Watts έχει το λόγο. Uh, I just Καταρχάς να πω ότι είναι πραγματικά πολύ πλούσια η συζήτηση που κάνουμε σήμερα. Και εγώ είμαι ηθοποιός και συγγραφέας και ποιήτρια, αλλά εδώ στο ε, κοινοβούλιο έμαθα την τέχνη του χαϊκού, σύντομες παρεμβάσεις. Είναι πολύ σημαντικό που ε, χρησιμοποιούμε την δημιουργικότητα και τον πολιτισμό στην ε, συζήτηση. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Ήθελα να ε, ευχαριστήσω τους εθελοντές για τη δουλειά που κάνουν, που πραγματικά πολλές φορές δημιουργούν πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες, τις οποίες μετά χρησιμοποιούν οι οργανώσεις, τα θεσμικά όργανα. Ας πούμε, ο Μάικλ Μάιερ που δημιούργησε μια, ένα ίδρυμα το, για την εβραϊκή κληρονομιά. Κάνει μια, ε, μια προσπάθεια χαρτογράφηση των συναγωγών στην Ευρώπη. Και ξέρω στην, στην Κρακοβία φέτο έγινε μια διάσκεψη για την αστική εβραϊκή κληρονομιά, στην οποία συμμετείχατε και ήταν κομμάτι των δραστηριοτήτων του προγράμματο του Ευρωπαϊκού Έτου. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικέ αυτέ οι δραστηριότητε, γιατί βλέπουμε ότι εκεί δουλεύει καλά η Ευρώπη και εκεί υπάρχουν πολύ καλέ πρακτικέ. Ένα σημείο θα ήθελα να τονίσω για την διατήρηση. Η αποκατάσταση καταστραμμένων έργων ίσως να μην μπορεί να γίνει στο μέλλον αν δεν χρησιμοποιήσουμε ψηφιακά εργαλεία. Ο σύρος που, έχει το, ε, που παρέχει το ίντερνετ στην Συρία δολοφονήθηκε. Πριν δολοφονηθεί τον είχε απαγάγει το ΆΙΣΕΣ και είχε δημιουργήσει, είχε δημιουργήσει μία ε, τρισδιάστατη απεικόνηση της Παλμύρας και χάρη σε αυτό θα μπορέσουμε στο, μέσο, στο μέλλον να δουλέψουμε πάνω στην αποκατάσταση. Αν δεν το ξέρετε, ψάξτε τη δουλειά του, είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικός. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε τώρα το Κοινοβούλιο του Κωσυφοπεδίου, αντιπρόεδρος της Επιτροπής α, ε, Πολιτισμού, Τόιτα Χάξη, Τέουτα Χάξη. Okay. Κυρίες και κύριοι, ε, σας καλώ να, να έλθετε στο Κωσυφοπαίδιο για να δείτε ποια από τις δύο ιστορίες που ακούσατε είναι η σωστή. Η δημοκρατία του Κωσυφοπαιδίου είναι έτοιμη να αναλάβει τι ευθύνε της έναντι της UNESCO και άλλων διεθνών οργανισμών. Κάτι το οποίο αμφισβητεί η Σερβία. Ζητούμε από τη Σερβία να μας επιστρέψει τα αρχεία και τα ε, πολιστικά αγαθά τα οποία κατέχει και ανήκουν σε εμά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε πάλι στον Βέσνερ Πεντικοβίτσο από το Κροατικό Κοινοβούλιο. Ε, Καταρχήν, ευχαριστώ που μου ξαναδίνετε το λόγο. Καταρχήν να πω ότι η Κροατία είναι μια χώρα με πολύ πλούσια πολιστική κληρονομιά, ενσώματη και άειλη. Έχουμε πολλές τοποθεσίες ε, αλλά και άειλη πολιστική κληρονομιά στην, που έχουν χαρακτηριστεί παγκόσμια πολιτική κληρονομιά από την UNESCO. Δυστυχώς ένα μέρος αυτών καταστράφηκε στον ε, πόλεμο της δεκαετίας του 90. Είχαμε πόλεις ολόκληρες που καταστράφηκαν διαρχείων του πολέμου. Πιο συγκεκριμένα το Ντουμπρόβνικ ή το Βούκοβαρ ήταν πόλεις που έπαθαν τεράστιες ζημιές, καθώς επίσης και το Ζάγκρεπ, η πρωτεύουσά μας. Σήμερα, 27 χρόνια μετά τον πόλεμο του 1993, το μεγαλύτερο μέρος ε, αυτών έχουν επισκευαστεί και συντηρηθεί χάρη και στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς επίσης και στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών. Είναι πολύ σημαντική η προστασία και η διατήρηση της πολιτικής κληρονομιάς, διότι μάλλον και εμείς ε, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους ε, διοργανώσαμε στο Ζάγκρεπ μια έκθεση ε, υπό την αιγίδα των κροατών συντηρητών, της οργάνωσης κροατών συντηρητών έργων τέχνης. Έκθεση η οποία τονίζει τη σημασία της συντήρησης και της προστασίας της πολιτικής κληρονομιάς. Ευχαριστώ. Ωραία. Πάμε τώρα στον Αντρέα Πόποβιτς. Επίσης ε, έχει ξαναπάρει το λόγο, αν θυμάμαι καλά, από το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου ξαναδίνετε το λόγο, που μου ξαναδίνετε την ευκαιρία να συνεχίσω με αυτά που προσπαθούσα να πω νωρίτερα. Δύο λόγια για την ε, πολιτιστική κληρονομιά του Μαυροβουνίου. η μεγαλύτερη πλειοψηφία των μνημείων μας είναι στο Κοτόρ, υπό την προστασία του UNESCO, από την ε, ενετική αλλά και την αυστρογγρική περίοδο. Επίσης έχουμε σημαντικό αριθμό εκκλησιών και μοναστηριών σε ένα αρκετά περιορισμένο χώρο με σημαντικό αριθμό μνημείων, χώρο περιορισμένο γεωγραφικά δηλαδή, το Κοτόρ ε, είναι ένας από τους παλαιότερους καθεδρικούς ε, ε, στην Ευρώπη από τον 9ο αιώνα Στη λίμνη Σκαντάρ επίσης έχουμε και στις όχθες της και σε νησάκια μέσα στη λίμνη σημαντικά μνημεία. Είναι μια περιοχή που είναι πραγματικά ο, ο πυρήνας ε, της μεσαιωνικής μας ε, παράδοσης. όπως και στα μοναστήρια της, του εσωτερικού της χώρας ε, που είναι μάρτυρες ε, της ε, τρικυμιώδους ε, ιστορικής πορείας της χώρας μας από τη Βυζαντινή περίοδο, αλλά και τυχογραφίες και φρέσκα πολύ σημαντικά. Ευχαριστώ. Και πάλι μέλος της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής Πολιτισμού, ο κύριος Στοβιέσκη. E, και πρόεδρε, Ε, ο συνάδελφός μου προηγουμένως μας ε, ένα πάρα πολύ όμορφο ποίημα. Ε, θα ήθελα και εγώ να πω δύο λόγια. Εκπροσωπώ το κοινοβουλίο μας. Ζητώ από την Κομισιό να μην είναι πολύ αυστηρή, να είναι πιο ευέλικτη σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση για, την, για τον πολιτισμό. Έχουμε δύο περιορισμούς. Αφενός γραφειοκρατικούς και αφετέρου το πεδίο των δράσεων οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Τα παραδείγματα που ακούσαμε ε, αυτές τις μέρες για αυτό το θέμα μας υποχρεώνουν να επιστρέψουμε σε αυτό και να το σκεφτούμε. Ευχαριστώ. Τελευταία ομιλήτρια για αυτό το πάνελ. Dragana Kostic από το Σερβικό Κοινοβούλιο. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να υπογραμμίσω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού ε, στη Σερβία έχει δεσμευθεί με προσπάθειες για να προστατεύσει το κληροδότημά μας, ε, το πολιτιστικό Έχουμε σημαντικές ε, παραδόσεις ε, ε, και έχουμε και σημαντική προέλευση της, της χριστιανικής παράδοσης με το σημείο γέννησης και του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Έχουμε σημαντικές δραστηριότητες επλαισίωσης της πολιτιστικής, τουριστικής μας οικονομίας. Τώρα, νομίζω ότι εδώ δεν είναι ο καλύτερος χώρος για να συζητήσουμε την ιστορία του κοσφοπεδίου, αλλά νομίζω ότι η αλήθεια θα προκύψει αργά ή γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε λοιπόν την ε, συζήτηση για το δεύτερο πάνελ και πάμε στο τρίτο πάνελ. Τελευταίο θεματικό πάνελ που ασχολήθηκε με τα θέματα της ε, πολιτιστικής κληρονομιάς και της εκπαίδευσης. Ήδη ακούσαμε βέβαια κάποια παρεμβάσεις σχετικά. Να δώσω τώρα το λόγο στην ε, Σαμπίνε Φερχάγεν, που ήταν η πρόεδρος χθες του θεματικού πάνελ, για να μας κάνει μια σύντομη ε, περίληψη. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Το πρώτο ε, τμήμα για την, της ε, περιείχε πολλές παρουσιάσει από την Κομισιόν για το τι έχει γίνει του τελευταίους 12 μήνε ε, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτου Πολιτιστική Συλλονομιάς. Για τα θέματα τη εκπαίδευση συγκεκριμένα, δύο συγκεκριμένα σχέδια έχει, ε, υπάρχουν στα πλαίσια αυτά. Ε, η διδαξικαλία των πολιτών για την πολιτιστική κληρονομιά και η χρήση τη πολιτιστική κληρονομιά ω εργαλείο για να μπορέσουμε να περάσουμε από, όλες, από όλους και από όλε τι ηλικίε εκπαίδευση θα συνεχίσει να παίζει το πολύ σημαντικό ρόλο σε διάφορα project τα οποία χρειάζονται πάρα πολύ σημαντική χρηματοδότηση. Η, με τη στήριξη των διαρθωτικών ταμείων και το Erasmus 2020 θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν ε, project πολιτιστικά, ε, το Discovery U, το Erasmus Plus επίσης αποτελούν ευκαιρίες για περαιτέρω συμμετοχή στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Υπάρχουν πολλά μακροπρόθεσμα project που έχουν προγραμματιστεί στα πλαίσια της πρόθεσης κληρονομιά. Η Κομισιόν έχει ένα σχέδιο δράσης εκπονήσει και υποστηρίζει διάφορε πρωτοβουλίε όπω η χειρονομιά στα σχολεία που έχει να κάνει και με την ηλεκτρονική ε, πλατφόρμα αδερφοποίηση, ε, με τα θέματα ε, εκπαιδευτικών και επίση προγράμματα από κοινού με την UNESCO και για την άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Ακούσαμε πολλέ παρεμβάσει από, από τα Εθνικά Κοινοβούλια για το πώ δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό. Το Ευρωπαϊκό Έτο Πολιτιστική Κληρονομιά πραγματικά κινητοποίησε την συμμετοχή και σε ευρωπαϊκό και σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Έγινε μεγάλη συζήτηση για το βασικά διδάγματα για τη μελλοντική δουλειά μα για την στήριξη των συνεργειών μεταξύ εκπαίδευση και ε, πολιτιστική κληρονομιάς. Είναι σημαντικό να εκτιμήσουμε την ε, ποικιλομορφία και τη άειλης και τη απτή πολιτιστική κληρονομιάς. Πρέπει να γίνουν περισσότερα για την προσβασιμότητα της πολιτιστική κληρονομιά. α πούμε, ε, με ζωντανέ παρουσιάσει που μπορούν να γίνουν και σε σχολεία και αλλού. Ε, είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι διάφορε ομάδε ε, εμπλεκομένων φορέων θα μπορέσουν να στηρίξουν τι κυβερνήσει. Η προσέγγιση από κάτω προ τα πάνω είναι πολύ σημαντική. Κυρίω το περιφερειακό επίπεδο μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Για την πολιτιστική κληρονομιά, για να μπορέσει να έχει αποτελέσματα για την εκπαίδευση, θα πρέπει να υπάρξει σωστό mainstreaming και στι ε, ακαδημαϊκέ συγκυκλίου. Η εκμάθηση τη πολιτιστική κληρονομιά θα πρέπει να ξεκινά το συντομότερο δυνατόν. Βεβαίω γίνονται διάφορα στον τομέα αυτό, αλλά πρέπει να ενισχυθούν. Η κινητικότητα επίση ε, των ε, επαγγελματιών μπορεί να βοηθήσει. Η ε, εξαποστάσεω εκμάθηση επίση. Η επίσημη τυπική εκπαίδευση μπορεί να συμπληρωθεί και από μη άτυπη εκπαίδευση και από σχετικές δράσεις και πρωτοβουλίες. Ο εθελοντισμό μπορεί να βοηθήσει επίσης για να διατηρηθεί η πολιτική κληρονομιά και να κινητοποιήσει την συμμετοχή σε προγράμματα τέτοια. Επίσης το, το Σώμα σε προσφέρει τέτοιε ε, ευκαιρίε μέσα σε ένα συγκεκριμένο ρυθμιζόμενο πλαίσιο. Και βεβαίω υπάρχουν και δυνατότητε εθελοντισμού των νέων, που είναι επίση εξίσου σημαντικέ. Σημαντικό είναι να ξεφύγουμε από την αποκλειστική στόχευση στι επιστήμε και να δώσουμε και στι τέχνε την ε, θέση που έχουν οι ε, τέχνες ε, δίνουν ένα κίνητρο στους νέους για να εμπλακούν, για να συμμετάσχουν, οπότε πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα και όχι ένα επιπρόσθετο μάθημα στα σχολεία. Οι τέχνες μπορούν να ε, βοηθήσουν επίσης και σε άλλα ακαδημαϊκά μαθήματα και ο σύνδεσμος πολιτισμού και εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικό και για την περαιτέρω εξέλιξη των βασικών ε, στοιχείων των προηγούμενων πάνελ της ε, ταυτότητα ας πούμε και τη αποκατάσταση. Αν δεν καταφέρουμε να έχουμε καλύτερη εκπαίδευση μέσω των ε, τεχνών και τη πολιτιστική κληρονομιάς θα χάσουμε την συνειδητοποίηση τη αξία τη πολιτιστική μα κληρονομιά. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. πλήρης η περίληψή σας. Από ό,τι φαίνεται ήταν πολύ ε, ενδιαφέρουσες οι συζητήσεις που κάνατε. Να δούμε τώρα τους ομιλητέ μας για αυτό το πάνελ. Ξεκινούμε με την Νικόλ Γκισε Κόνιγκ. Είναι ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο ULB εδώ στις Βρυξέλλες και θα μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση. Σας ακούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αγαπητοί συμμετέχοντες. Ζητήθηκε μια μελέτη για τις συνέργειες μεταξύ των πολιτικών πολιτισμού και ε, παιδείας για να έχουμε πιο αποτελεσματική συνεργασία προκειμένου να ενισχύσουμε την δυνατότητα των πολιτών όχι μόνο να συμμετέχουν αλλά και να συμμετέχουν υπεύθυνα. Υπάρχει μεγάλη σύγχυση ε, και γλωσσική μεταξύ άλλων για το τι σημαίνει εκπαίδευση στον πολιτισμό, εκπαίδευση στην ε, πολιτιστική παράδοση και κληρονομιά, ε, η πολυμορφία των φορέων και των σωμάτων που ασχολούνται με τις ε, θεματικές αυτές ε, ε, σχετίζονται με το θέμα αυτό. Υπάρχουν συνέργειες όμως. Η αδελφοποίηση πόλεων στις οποίες, στην οποία προχωρούμε τελευταίο. Πολλές άλλες πρωτοβουλίες όπως το το όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη, οι υπόγειες, ε, ε, οι υποθαλάσσιες πόλεις κτλ. Ε, σκεπτόμαστε το μέλλον ε, και της κληρονομιάς αυτής, του κληροτήματος αυτού και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα ακόμα που μπορούμε να αναφέρουμε, αλλά οι συνέργειες αυτές είναι ανεπαρκείς. Πολύ συχνά βλέπ, είναι αντιληπτή η δραστηριότητα αυτή ε, ως μεμονωμένες πρωτοβουλίες που δεν είναι συνδεδεμένες με, με, πια πιο, με, με, πια πιο, μια πιο μακροπρόθεσμη προσπάθεια, πιο διαρθρωμένη δηλαδή προσπάθεια για να δούμε τι σχεδιάζουμε για το μέλλον ε, στα, δια, στα πλαίσια των διαφορών έργων ώστε να επαναφέρουμε ε, μεταξύ άλλων και απασχόληση και διαρθρωτικές βελτιώσεις στα σχολικά προγράμματα. Οι συνέργειες δεν είναι δομικά ενσωματωμένες στα συστήματα παιδείας μας. Πρόσθετες συστάσεις και μελέτες αναφέρονται και πολύ συχνά θα παραπέμπουμε σε αυτές σχετικά με την παιδεία θα συστήναμε προς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υλοποιήσουν τις ακόλουθες συστάσεις μέσω των καταλήλων ευρωπαϊκών πολιτικών. Να, να ενθαρρύνουν την ενσωμάτωση σε όλα τα σχολικά προγράμματα και επίσημης και άτυπης μάθησης, να έχουμε σαφείς ορισμούς σχετικά με τον πολιτισμό, την πολιτιστική παράδοση, την ε, εκπαίδευση, την εκπαίδευση στην τέχνη και στον πολιτισμό και στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού γλωσσαρίου. Να επιτρέψουμε καλύτερη διάχυση βελτίστων πρακτικών και παραδείγματα εκμάθησης από αγαθά πολιτιστικά, διαβίου μάθηση, την βέλτιστη πρακτική της Επιτροπής Πολιτισμού του Διεθνού Συμβουλίου των Μουσείων και κοινέ πληροφορίες, κοινά δεδομένα εξασφαλίζοντας ότι θα έχουμε διαρκώς επικαιροποιημένους ε, συνδέσμους μεταξύ των τομέων του πολιτισμού και της παιδείας, αποφεύγοντας υπερβολική ενημέρωση που πολύ συχνά σκοτώνει τη γνώση. Χρειαζόμαστε ευαισθητοποίηση σχετικά με την κληρονομιά, μέσω της χρησιμοποίηση του Erasmus Plus, ε, των προγραμμάτων διαβίου μαθήσεως και άλλων προγραμμάτων των συναρμοδίων φορέων. Και βέβαια η χρηματοδοτική πόρη που θα είναι απαραίτητη μακροπρόθεσμα. Αυτό που ήδη αποδείχθηκε χρήσιμο είναι να έχουμε συνέργειες μεταξύ των διαφόρων αρμοδίων επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί να πολλαπλασιάζουμε εκδηλώσεις μεμονωμένες. Ja, vielen herzlichen Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Το τελευταίο βεβαίως έχει να κάνει και με τις ε, διαπραγματεύσεις που κατέρευσαν για τον ε, προϋπολογισμό. Ε, όντως πρέπει λίγο πιο βιώσιμα να εφαρμόζουμε τους, να εκτελούμε τους ε, προϋπολογισμούς, όταν βεβαίως τους έχουμε, όταν έχουμε τα κονδύλια. Λοιπόν, Ραφαέλ Ζεράρ από την Γαλλική Εθνοσυνέλευση να ζητήσω να πάρει το λόγο τώρα, γιατί θέλει να φύγει πιο νωρίς, οπότε θα του δώσουμε τώρα το λόγο και οι υπόλοιποι θα παρέμβετε αργότερα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί βουλευτές, εκπροσωπώ την Επιτροπή Πολιστικών Θεμάτων της ε, ε, Γαλλικής Εθνοβουλής. Εθνοσυνέλευση, συγγνώμη. Μιλάμε για την πολιστική κληρονομιά, ε, κτίρια αλλά και μουσική, ζωγραφική κλπ. Όλα αυτά είναι κομμάτια των προηγούμενων γενιών που δεν είναι δυνατόν να τα περάσουν στις επόμενες γενιές χωρίς τη βοήθεια της εκπαίδευσης. Η Ευρώπη πάντοτε χαρακτηριζόταν από κινήματα αρχιτεκτονικά και άλλα οι, που υπερεύαιναν τα σύνορα και τις αυτοκρατορίες από την αρχαία ελληνική εποχή, τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία κλπ. μέχρι σήμερα. Η, η αρχιτεκτονική, για παράδειγμα, έχει δημιουργήσει ένα κοινό περιβάλλον σε όλη την ε, Ήπειρο, κάτι που μας οδηγεί στο να νιώθουμε πως ανήκουμε σε κάτι υπερεθνικό. Οπότε η πολιτική δεν θα πρέπει απλώ να διατηρείται αλλά και να μεταδίδεται σε επόμενες γενιάς, γενιές. Ε, μέσω αυτού οι νέοι θα πρέπει να μαθαίνουν το διάλογο ε, και τη συμβίωση. Είχε πάει στο Μόλεμπεκ ο πρόεδρο Μακρό και είχε πει τότε στους νέους ότι θα πρέπει να ορίζουν τον εαυτό τους όχι μόνο μέσω τη γειτονιά τους αλλά και μέσω της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το αίσθημα του ανήκει περνάει μέσα από τι οικονομικές ανταλλαγές βέβαια αλλά κυρίως μέσα από τι πολιτιστικέ και εκπαιδευτικέ ανταλλαγέ. Για να διευκολύνουμε αυτέ τι ανταλλαγέ όπω και η Πορτογαλία Έχουμε αποφασίσει ε, την εκμάθηση της μιας πρώτης ξένης γλώσσας από το δημοτικό σχολείο, από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης ε, θέλουμε η πολιστική δημιουργία να φτάσει σε όλους τους ε, μαθητές ανεξαρτήτως της προέλευσής τους κοινωνικής ή άλλης. Στο τέλος του προηγούμενου έτους ε, δημοσίευσαμε ένα σχέδιο που θα επιτρέψει όλους του μαθητές από τα 3 μέχρι τα 18 ε, έτη να ακολουθούν μια εκπαιδευτική πολιτιστική διαδρομή πλήρη. Όχι πως ε, αυτό έλειπε παλιότερα, έχουμε πολλά μαθήματα τεχνών στα σχολεία, τώρα απλώς θέλουμε μια πιο συνολική σφαιρική καλλιτεχνική προσέγγιση, όχι μόνο μέσω της μουσικής, της ζωγραφικής, αλλά και μέσω της αναζήτησης και της χρήσης των αντικειμένων. Αυτή τη στιγμή το, από εδώ και πέρα το 10% του εκπαιδευτικού χρόνου θα αφιερώνεται στην, στις καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Επίσης, εξωσχολικές δραστηριότητες θα προτείνονται στους μαθητές από, την, από το ε, από την προσχολική εκπαίδευση, από τα τρία χρόνια της ζωής, από τον τρίτο χρόνο ζωής των παιδιών μας. Ε, δίνουμε ιδιαίτερη, ιδιαίτερο βάρος στη μουσική που θα διδάσκεται σε όλα τα σχολεία. Εισαγωγή στη μουσική και από το Σεπτέμβριο του 2018 ε, δημιουργήσαμε ένα σύστημα που οι παλιότεροι μαθητές δίνουν συναυλίες και υποδέχονται έτσι τους καινούριου μαθητές. Ιδιαίτερα ε, στα πιο προβλημα... στις πιο προβληματικές ε, γειτονιές, ε, κάνουμε παρεμβάσεις στα σχολεία. Επίσης είναι πολύ σημαντική η αρχιτεκτονική, διότι έχει σχέση με τον τρόπο ζωής των πολιτών μας. Το καλλιτεχνικό λοιπόν πρόγραμμα προβλέπει μία τουλάχιστον επίσκεψη κατέτος σε ένα αρχιτεκτονικό έργο. Αυτό επιτρέπει στους μαθητές να προετοιμαστούν για το μέλλον, για την καλλιτεχνική τους εκπαίδευση στο μέλλον. Οι νέοι για ένα χρόνο θα έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν μία από τις εμπειρίες που τους ενδιαφέρει μέσω ενός πολιτιστικού πάσου, όπως το λέμε, έτσι ώστε να ασχοληθούν πιο ε, βαθιά με αυτό που τους ενδιαφέρει. Ψηφιοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι ότι ε, βοηθάει τους νέους. Αυτή τη στιγμή τους δίνουμε μια επιταγή 500 ευρώ το χρόνο, bonus κουλτούρα το ονομάζουμε. Η χρήση αυτών των 500 ευρώ ε, θα γίνει ε, με πιο αυστηρούς όρους από ό,τι γίνεται στην Ιταλία, αν και εμπνευστήκαμε εμείς από την Ιταλία. Ίσως είναι ένα σύστημα το οποίο θα έπρεπε να διευρυνθεί, ίσως όχι με χρηματικές φορές, αλλά με ε, ένα τρόπο λιγότερο οικονομικό, που θα, χρηματικό μάλλον, που θα έσπρωχνε τους ε, μαθητές να έρθουν σε επαφή με τα πολιτικά αγαθά όλων των χρόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά θετικά παραδείγματα μας αναφέρατε. Ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στην Μαρία Αουγκούστα Σάντος από το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο. Σας ακούμε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ ονόματος της ε, Πορτογαλικής Βουλής σας χαιρετώ, χαιρετίζω όλους και όλες. Είμαστε η μνήμη που έχουμε και οι ευθύνε που αναλαμβάνουμε. Χωρί μνήμη δεν υπάρχουμε. χωρί ευθύνη ίσω δεν αξίζουμε να υπάρχουμε. Αυτά τα έγραψε ο Ζωζέ Σαραμάγκου που έχει ε, πάρει το, κερδίσει το βραβείο Νόμπελ ε, στη λογοτεχνία. Το, Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτικής Κληρονομιάς είναι η αναγνώριση της κοινή μας ε, μνήμης και η ανάληψη της ευθύνης για την ανάδειξη της μνήμης. Ε, ταυτόχρονα όμως είναι και η οθέτηση ε, μιας εκπαίδευσης και μιας επιστήμης ως ε, δρόμους για την γνώση του, του παρελθόντων μας. Είναι η κοινή μας κληρονομιά αλλά είναι και η ζωή που θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές. Η Πορτογαλία είναι ανοιχτή στον κόσμο, έχει μια ιστορία και μια διασπορά σε όλες τις υπήρους. Είναι μια χώρα ανοιχτή και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μια χώρα που ε, θέλει η εκπαίδευσή της να, είναι, να, μην, είναι χωρίς αποκλισμούς, να ενισχύσει τον αλφαβητισμό και το αίσθημα του πολίτη. Με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι η κουλτούρα είναι πυλώνας της δημοκρατίας και της εθνικής ταυτότητας. Από το Σύνταγμά μας προβλέπεται η δημοκρατική πρόσβαση στη δημιουργία και την απόλευση των πολιτικών αγαθών. Αυτό μας υποχρεώνει να διατηρούμε, να ανακτούμε και να διαδίδουμε την πολιτική μας κληρονομιά μέσω μιας πολιτιστικής πολιτικής οριζόντιας ιδιαίτερα μέσω της επιστήμης και της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση απαιτεί μια μεθοδική και μόνιμη εργασία. Γι' αυτό το λόγο η ενίσχυση των τεχνών ε, και των ανθρωπιστικών σπουδών είναι απολύτως απαραίτητη. Η κινητοποίηση της έρευνας και της επιστήμης μαζί με την ενίσχυση της χρήσης των νέων τεχνολογιών και της ψηφιοποίησης του πολιστικού περιεχομένου αποτελούν δράσεις προτεραιότητας για την ανάδειξη και την ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής μας ταυτότητας. Επίσης συνεισφέρουν προκειμένου να εμβαθυνθεί ο εκδημοκρατισμός της πρόσβασης στον πολιτισμό εκ μέρους όλων. Θα έπρεπε αυτό να είναι παγκόσμιο καθολικό δικαίωμα. Η ανάδειξη της, ε, του πολιτισμού ε, περιλαμβάνει πολλές δράσεις και διάφορα σχέδια ιδιαιτέρως μέσω της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου για τις Τέχνες για τους μαθητές των σχολείων, όπως έχει γίνει στο παρελθόν με το Εθνικό Σχέδιο Ανάγνωσης και το Εθνικό Πρόγραμμα Κινηματογράφου. Αυτό μας οδηγεί στο να εργαστούμε σε δίκτυο, σε συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, καθώς επίσης και με την κοινωνία των πολιτών. Το πολιστικό η πολιστική κληρονομιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κοινή μας ταυτότητα. Είναι η ευρωπαϊκή ταυτότητα. Είναι η ε, ε κομμάτι του τριγώνου που αποτελούν η εκπαίδευση και η επιστήμη, ο πολίτης και η πολιστική κληρονομιά. η εκπαίδευση είναι ένας ε, παράγοντας ανάπτυξης οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής. Και όπως αναγνωρίζεται από την UNESCO, η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι ε, να κινείται προς την κατεύθυνση α, της α, ε, κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας. Στην, στην εκπαίδευση θα πρέπει να μην γίνονται εξαιρέσει, να είναι ισότιμοι για όλους και να βοηθήσει τους μαθητές να ε, εντάσσουν στην καθημερινή του ζωή τις αξίες και τον πολιτισμό. Είναι πολύ σημαντικές οι συνέργειες. Υπάρχουν, αλλά δεν είναι αρκετές. Ούτε και είναι αρκετά διαρθρωμένες, έτσι ώστε να γίνουν πιο σημαντικές, για την, πιο χρήσιμες για την εκπαίδευση. Χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία, χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία. Χρειαζόμαστε, χρειάζεται να είμαστε ικανοί να εμβαθύνουμε σε αυτή τη συνεργασία, για την οποία ε, θα πρέπει να μοιραστούμε γνώση, να μοιραστούμε αξίες και πόρους. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης δεν υπάρχουν πια κουλτούρες κλειστές. Αυτή τη στιγμή βασιζόμαστε σε ένα πολιτικό διάλογο στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κλείνουν 70 χρόνια από την δήλωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 40 χρόνια από την υπογραφή από την Πορτογαλία της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Ευρώπη πρέπει να γίνει ένας φάρος πολιτιστικός και εκπαιδευτικός. Γιατί ο πολιτισμός μας εξανθρωπίζει. Η Ευρώπη δεν χρειάζονταν ποτέ πιο πολύ δράση, πολιτική δράση, πιο ανθρωπιστική δράση. Τώρα είναι μεγαλύτερη αυτή η ανάγκη. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια κοινή πολιτιστική κληρονομιά με ελευθερία. Ο Καμίους είχε γράψει «Χωρίς την κουλτούρα και την αντίστοιχη ελευθερία, η κοινωνία, όσο τέλεια και να είναι, δεν πάβει να είναι ζούγκλα. Γι' αυτό το λόγο η αυθεντική δημιουργία είναι δώρο για το μέλλον. Ευχαριστώ. Σα vielen, vielen herzlichen Dank. Σας ευχαριστώ πολύ για την παθιασμένη σας παρέμβαση. Προχωρούμε με την Τεούτα Χάξιο από το Κοινοβούλιο του Κοσφοπεδίου. Thank you. We... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ε, συμφωνήσαμε ότι εγώ ε, εξ ονόματος όλης της ομάδας θα πω δύο λόγια για αυτό, υπό αυτό το σημείο μάλλον. φίλοι, η πολιτιστική κληρονομιά του Κωσυφοπεδίου είναι πολύ πλούσια και ξεκινάει από τα αρχαία χρόνια. Εμείς πιστεύουμε ότι η ποικιλότητα, η διαφορετικότητα της ε, πολιτιστικής κληρονομιάς είναι κάτι πολύτιμο και πρέπει να το προστατεύσουμε. Το προστατεύουμε λοιπόν υπό το Σύνταγμα και υπό την νομοθεσία μας. Εμείς επενδύουμε στην πολιτιστική παράδοση και κληρονομιά όλων των κοινοτήτων ισότιμα και με την πλούσια πολιτιστική παράδοση που έχουμε είναι πολύ καλό καθότι είναι και τμήμα της ευρωπαϊκής κληρονομιάς η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεισφέρει, να επενδύσει και αυτή στην προστασία τους. Η πραγματικότητα είναι πολύ μακρινή από αυτά που ακούσαμε ε, σήμερα από τους εκπροσώπους ε, της Σερβίας. Ε, έχουν αφαιρέσει πολλά τεμάχια, πολλά αγαθά πολιτιστικά από τη χώρα μας και πρέπει να μας επιστρεφούν. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα στον Αμρουλά Ισλέρ Καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη που σήμερα είχαμε ένα πρόβλημα με την τουρκική διερμηνία. Ε, θα ψάξουμε γιατί έγινε, αλλά πραγματικά ε, εγώ είμαι πολύ εκνευρισμένη. Χτες τα είχαμε καταφέρει. Ε, δυστυχώς πρέπει να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί σήμερα δεν καταφέραμε να έχετε τουρκική διερμηνία, αλλά ξέρω ότι έχετε προετοιμάσει στα αγγλικά την παρέμβασή σας, οπότε σας δίνω το λόγο για να μας την παρουσιάσετε. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη διοργάνωση της σημερινής συζήτησης. Η ανταλλαγή γνώσεων εδώ σίγουρα θα συνεισφέρει στην περαιτέρω οικοδόμηση των σχέσεών μας έχουμε την τελική φιλοδοξία να γίνουμε πλήρες μέλος και δίνουμε και εμείς πολύ μεγάλη σημασία στα θέματα της πολιτικής, πολιτιστικής κληρονομιάς και της ε, παιδείας. Εντός του κεφαλαίου λοιπόν 26 αυτού ε, συνεργαζόμαστε σε μια ευθυγράμμιση προς τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τεχνικά είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις υπό το κεφάλαιο αυτό. Δυστυχώς όμως έχουμε τεχνητά εμπόδια και μπλοκάρισμα της προόδου των συζητήσεων. Η ανάπτυξη των πολιτικών που αφορούν στον πολιτισμό και την παιδεία ή την προαγωγή της ε, πολιτιστικής ποικιλότητα και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι πολύ σημαντικές. Εμείς συμμετέχουμε στον Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τον Πολιτισμό και τις βελτιώσεις ε, της διεθνούς συνεργασίας, ιδιαίτερα με την UNESCO. Εμείς είμαστε μέρος, συνυπογράφουμε πάρα πολλές διεθνείς συμβάσεις ε, ε, σχετικά με τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά. Από το 2004 συμμετέχουμε σε προγράμματα υποστήριξης ε, πολιτιστικά και εκπαιδευτικά στο πλαίσιο των οποίων προγραμμάτων ε, μεταφράζονται πολύ σημαντικά κείμενα, αν καταλάβαμε καλά τον ομιλητή, και έχουμε και πολύ ενδιαφέροντα έργα διεθνούς συνεργασίας. Συνεργαζόμαστε με την UNESCO, την Interpol και τον Διεθνή Οργανισμό Τελωνίων για την αποτροπή του λαθρεμπορίου κοιμηλίων και αγαθών της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τέχνης και να επιστραφούν τα στοιχεία αυτά στη χώρα προέλευσής τους. Συμμετέχουμε σε όλες τις σημαντικές διεθνείς συμφωνίες προστασίας των αγαθών του πολιτισμού και της τέχνης ως χώρα προορισμού θα πρέπει επίσης να συμμετέχουμε επικοδομητικά. Όλες οι χώρες πρέπει να ε, εντείνουν τις προσπάθειές τους, τη συνεργασία τους και να αντιληφθούν τις ευθύνες που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις. Εμείς καταδικάζουμε έντονα την καταστροφή ε, πολιτιστικών αγαθών και μνημείων πρέπει οπωσδήποτε να αποτρέπουμε την διεθνή λαθρεμπορία αγαθών πολιτιστικής κληρονομιάς και τέχνης και θα πρέπει να επιστραφούν όλα τα κλαμμένα αυτά ευρήματα στην, στις ε, χώρες από τις οποίες προέρχονται. Διοργανώσαμε εργαστήρια και για τους δικούς μας υπευθύνους ε, επιβολής του νόμου και προγράμματα ευαισθητοποίησης για όλους τους συναρμοδίους ε, κρατικούς φορείς και προσπαθούμε να συνεργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή και με τις γειτονικέ μας χώρες. Έχουμε αναλάβει επίσης νέα νομικά μέτρα σύμφωνα προς τις διατάξεις για την προστασία της πολιτικής κληρονομιάς και συμμετέχουμε και σε διάφορα προγράμματα και κατάρτισης και εκπαίδευσης Προγράμματα επίσης διαβίου μαθήσεως που είναι πάρα πολύ σημαντικά για τους νέους και τους φοιτητές. Θα ήθελα να κλείσω αγαπητοί συνάδελφοι υπογραμμίζοντας το εξής. Ο πολιτισμός μας, η θρησκεία μας, η κοινωνική μας παράδοση δεν μας επιτρέπουν να καταστρέφουμε μνημεία τέχνης και πολιτιστικής παράδοσης. Υπό την Οθωμανική περίοδο είχαμε κέντρα ειρήνης και συνύπαρξης ανταυτών σήμερα μετά την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας βλέπουμε την καταστροφή που υφίστανται πάρα πολλά θρησκευτικά κέντρα και μνημεία λόγω του αυξανόμενου εθνικισμού. εμείς δεσμευόμαστε να, προστατευτούμε, να προστατεύσουμε όλα τα θρησκευτικά κτίρια, ναούς, μνημεία λατρείας όλων των θρησκειών. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της σημερινής συζήτησης. Ευχαριστώ. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und man kann nur hoffen, wenn das vielleicht auch politisch... Ευχαριστώ. Όντως ε, είναι σημαντικό να είμαστε σε επαφή με την Τουρκία. Καμιά φορά ο διάλογος ε, συναντά κόμματα, αλλά ίσως ε, στον τομέα του πολιτισμού να τα έχουμε καταφέρει λίγο καλύτερα. Ευχαριστώ λοιπόν που σήμερα έχετε, είστε εδώ και παίρνετε μέρος στην ε, σημερινή μας διάσκεψη. Λοιπόν, έχουμε τώρα μέχρι και τέταρτο έχουμε χρόνο για συζήτηση. Θα προσπαθήσω όσο το δυνατόν περισσότεροι να λάβετε το λόγο, αλλά πάλι θα σας διακόπτω. Ξεκινούμε με την Μαρή Λουίζ Οντόνελ από την Γερουσία της Ιρλανδίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πρόεδρε, ρωτήσατε για την, ε, ταυτότητα, κρίση, για την κρίση ταυτότητας. Ποιοι είμαστε, πού είμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Θα πρέπει να απαντήσουμε τα ερωτήματα αυτά, αν δούμε την ε, κρίση της ε, ταυτότητας και αν δούμε την ε, αξιοπρέπεια, την γλώσσα, τη γνώμη, είναι η δύναμη των τεχνών, της μουσικής, των οπτικοακουστικών τεχνών της λογοτεχνίας και της, πίεσης, και της πίεσης Αυτή είναι η δύναμη που έχουμε εμείς στα χέρια μας μέσω της εκπαίδευσης, γιατί αν, δείτε την πραγματική ε, ισχύ, βρίσκεται στην πνευματική, ε, στο, στο πνεύμα, στην, ε, στο σημείο που ανήκουμε, στην αίσθηση του ανήκειν, γιατί σίγουρα δεν θα, δεν θα προσπαθήσω εγώ να, μέσω της άλγευρας να βρω προ, λύσεις στα προβλήματά μου, γιατί λοιπόν οι τέχνες βρίσκονται στο, στο επίκεντρο γιατί δεν βρίσκονται μπροστά στο, στα προγράμματα STEAM και είναι κάπου στο τέλος. Γιατί βρίσκονται μέσα σε ένα γενικότερο πολιτιστικό πεδίο, γιατί δεν μπορούμε να τα πούμε ξεκάθαρα, ρητά και κατηγορηματικά. Γιατί σε όλα όσα έχουμε αναφέρει σήμερα, όλες αυτές οι πτυχές των τεχνών ήταν ε, οι ε, παγωγικές προς την ε, ισχύ και την δύναμή τους. Αναφέραμε πολλές, πολλά παραδείγματα. Κάθε φορά που ανοίγω την ε, τηλεόραση εγώ βλέπω τραπεζίτες να μιλάνε για λεφτά, από πού θα τα πάρουν, πού θα τα δώσουν. Και πραγματικά τα αποτελέσματά τους είναι καταστροφικά. Θέλουμε να υπάρχει η ίδια δύναμη όπως έχουν οι τραπεζίτε τραπεζίτες με αυτή που έχουν την, ε, με τους ε, καλλιτέχνες. Γιατί είναι η πραγματικά α, πνευματική δύναμη και είναι η πνευματική οικονομία που πρέπει να προωθήσουμε. Ευχαριστούμε για την παθιασμένη παρέμβαση. Νομίζω συμμεριζόμαστε όλοι χωρίς καμία αμφιβολία και αντίθεση. Άννα Βασιλεύσκα τώρα, από την ε, Πολωνική Γερουσία που είστε. Παρακαλώ, ένα λεπτό στη διάθεση σας έχετε. Ε, ε, Ευχαριστώ. Εκπροσωπώ το Πολωνικό Κοινοβούλιο και εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού. Να σας μιλήσω για τις δικές μου σκέψεις. Πράγματι η εκπαίδευση πρέπει να βασίζεται στην πολιτική κληρονομιά. Είναι δύο πυλώνες του ίδιου πράγματος, έχουν τα, τους ίδιους στόχους κατά βάση. Και το ένα πρέπει να εμπνέεται από το άλλο. Πολιτική κληρονομιά από την εκπαίδευση και το αντίστροφο. Η γνώση της πολιτικής κληρονομιάς θα πρέπει να ξεκινάει από πολύ νωρίς στη ζωή των παιδιών από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα έλεγα. Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Η πολιτική κληρονομιά θα πρέπει να είναι προσβάσιμη και μάλιστα με τρόπο που να εμπνέει και να ενδιαφέρει τα παιδιά. Μέσω παιχνιδιών ή άλλου διδακτικού υλικού. Ε, μέσω της ε, ψηφιακής τεχνολογίας επίσης ε, μπορούσε, θα μπορούσαν τα παιδιά να βλέπουν πώς ήταν τα αρχαία μνημεία πριν και πώς είναι τώρα. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά συνδέονται τόσο με τη σημερινή πραγματικότητα όσο και με το παρελθόν τους. Η εκπαίδευση, στη δευτερο... η... η δευτεροβάθμια εκπαίδευση επίσης είναι πολύ σημαντική για την προστασία Τη πολιτική οικονομίας και για την προώθηση μια κοινή ταυτότητα. Οι τοπικέ κουλτούρε επίσης θα πρέπει να προαχθούν μέσω της ενημέρωσης και των δασκάλων και των καθηγητών. Ευχαριστώ. Πάλι μέλος της ε, δικής μας Επιτροπής. Ένα λεπτό. Να πω ότι η εκπαίδευση πρέπει να ισχύει και για εμάς. Και εμείς πρέπει να μάθουμε. Και εμείς πρέπει να είμαστε αρκετά ταπεινοί ώστε να παραδεχτούμε ότι δεν ξέρουμε τα πάντα και να εμπλακούμε σε πολύ βασικές δραστηριότητες. Εγώ χαίρομαι που έχουμε ε, σύνδεση με το δίκτυο για τα μουσεία και πήγαμε στο Μάστριχτ για μια επίσκεψη. Υπάρχει και ένα σχετικό φιλμ. Σας ε, ζητώ να το δείτε, αλλά μπορείτε και εσείς να κάνετε μια δική σας ε, μαθητεία, ας πούμε, στα τοπικά σας μουσεία. Οπότε μπορείτε και εσείς να δουλέψετε πίσω από, από το παρασκήνιο, να δείτε πώς δουλεύουν οι οργανώσεις αυτές και ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Και σίγουρα θα μπορέσουμε να υπερασπιστούμε πολύ καλύτερα έτσι τα συμφέροντα του κλάδου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σεβαστάκης έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, στην πόλη μου, την Αθήνα, στην πατρίδα μου, την Ελλάδα, σε κάθε έργο, σε κάθε εξκαφή ανακαλύπτονται αρχαία ε, υπολείμματα ενός πολιτιστικού αποθέματος, που σημαίνει ότι ο πολιτισμός του παρελθόντος σχετίζεται με τον αστικό σχεδιασμό το σύγχρονο, σχετίζεται με την πολεοδομία, σχετίζεται με την χωροταξία, σχετίζεται με την πρόσληψη της φύσης. Επομένως, η περιπατητική εμπειρία, η εμπειρία στην πόλη, η εμπειρία στη φύση αποτελεί μια μορφή εκπαιδευτικού γεγονότος. Η ίδια η πρόσληψη του παρελθόντος από το σύγχρονο θεατή είναι εκπαιδευτικό γεγονός. Εν οι μεγάλες πιέσεις με τις μετακινήσεις πληθυσμών δημιουργούν μια γενικότερη πολιτιστική ανασφάλεια. Επομένως, η πρόσληψη της τέχνης του παρελθόντος του πολιτιστικού αποθέματος συσχετίζεται με αυτή την δομική πολιτιστική ανασφάλεια του σύγχρονου αναγνώστη. Αυτό εγώ θα ήθελα να καταθέσω, να το βάλουμε μέσα στη συζήτηση. Το πρόβλημά μας δεν είναι να διασώσουμε μόνο με τεχνικούς ή τεχνολογικούς τρόπους ή με αναπαραστάσεις που τα σύγχρονα μέσα μας ε, εξασφαλίζουν το παρελθόν μας μόνο, αλλά να μπορέσουμε να έχουμε έναν ενεργό, ανοιχτό οφθαλμό, ένα σύγχρονο μάτι που θα μπορεί άφοβα να το παραλάβει και με αυτόν τον τρόπο να συνδέσει τη νέα ενότητα που έχει ανάγκη η Ευρώπη. Vielen herzlichen Dank. Madame Ευχαριστώ. Η κυρία Μπίλτ. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρωτοβουλία υπαριθμών 4 αφορά στην πολιτική κληρονομιά σε μετάβαση, ιδιαίτερα ε, την θρησκευτική κληρονομιά, ε, που είναι πολύ σημαντικό θέμα στην χώρα μας, όπως με επαναχρήσεις εκκλησιών, στον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης για παράδειγμα, Πρέπει λοιπόν να υποστηρίζουμε τις θρησκευτικέ κοινότητες, τις τοπικές. Ε, στο Κωσυφοπαίδιο υπάρχει μια πολύ σημαντική ε, ε, ορθόδοξη παράδοξη για τους Σέρβους, αλλά και σήμερα το πρωί είχαμε επίθεση σε δύο λεωφορεία προσκυνητών ή στην περιοχή. Πώς μπορούμε λοιπόν να προστατεύσουμε την πολιτική μας κληρονομιά εάν δεν σεβόμαστε τα ίδια τα μνημεία, τα ίδια τα κτίρια. Είναι ένα θέμα παιδείας και πολιτισμού. Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Λουίτζι Γκάλο από το Ιταλικό Κοινοβούλιο και μετά πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή τη συζήτηση. Θα χρησιμοποιήσω αυτό το λεπτό για να αναφερθώ και εγώ ε, στο άρθρο 175 και τα θέματα πολιτισμού και παιδείας. Το άρθρο λοιπόν 175 λέει ότι πρέπει να αναπτύξουμε την ευρωπαϊκή διάσταση της παιδείας. Αυτό θα σήμαινε και να έχουμε ένα παιδαγωγικό πρότυπο κοινό από την ιστορία των χωρών μας να βρίσκει μια κοινή ταυτότητα. Άκουσα αρκετές παρεμβάσεις για το πώς θα μπορούσαμε να έχουμε μια εμβάθυνση στο πολιτιστικό πεδίο και ε, η αυτή η εμβάθυνση δεν μπορεί παρά να επιτευχθεί μέσω της επίσκεψης στους ε, τόπους, τους αρχαιολογικούς χώρους, τους χώρους της πολιτιστικής κληρονομιάς, την, ε, συμμετοχή της έρευνας και όταν αναπτύξαμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, εμείς τουλάχιστον στην Ιταλία ε, ε, υπογραμμίσαμε το θέμα της ε, κατάρτισης και της εκπαίδευσης των καθηγητών πανεπιστημίου, που είναι ακαθίσταται όλο και πιο σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την τελευταία παρέμβαση. παθιασμένη σε παρεμβάσει σήμερα, αλλά δεν πρέπει να το παρεξηγούμε. Είναι πράγματα που μας απασχολούν ε, πολύ. Ο πολιτισμός και η εκπαίδευση ε, είναι θέματα σημαντικά, δεν πρέπει να τα ξεχνούμε. Λοιπόν, μπορούμε να περάσουμε στο τέλος τώρα, στο τελευταίο κομμάτι της ε, διάσκεψής μας με την παρουσία του Επιτρόπου Ναύρατσιτς, Επιτρόπου για την Εκπαίδευση. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ και ευχαρίστως να σας δώσω το λόγο για να κάνετε την παρουσίασή σα για να κλείσετε κιόλα πρακτικά τη σημερινή διάσκεψη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αυτές οι δύο τελευταίες μέρες ε, αποτέλεσαν ε, μία στιγμή για στοχασμό. Να σκεφτούμε σημεία σημαντικά που άπτονται της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ήταν μια στιγμή να δούμε το ευρωπαϊκό μέλλον, όπου η πολιτιστική κληρονομιά θα παίζει σημαντικό ρόλο και θα υποστηρίζετε ακόμη καλύτερα για να συζητήσουμε πώς μπορούμε από κοινού αυτό το όραμα να γίνει πραγματικότητα. Είναι επίσης μια στιγμή και για μένα για να σας ευχαριστήσω που υποστηρίξατε αυτή την υπέροχη πρωτοβουλία. Ήδη από το 2017 η στήριξή σας ήταν θεμελιώδος σημασία ώστε να περάσει η απόφαση αυτή για το ευρωπαϊκό έτος. Και μετά ε, μπορέσαμε να καταλήξουμε και στον προπολογισμό. Το 2018 η στήριξή σας παρέμεινε αταλάντευτη όταν ξεκίνησαν τα διάφορα project σε όλη την Ευρώπη. Προωθήσατε τον, το ευρωπαϊκό έτος και στους συναδέλφους σας και στις γειτονικές σας χώρες. Μπήκατε στο δίκτυο της και στην Επιτροπή των Εμπλεκόμενων Φορέων και των Συντονιστών και κυρίως φέρατε το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Χρονομιάς στις ζωές των ε, πολιτών σας. 11.500 ε, δραστηριότητες διοργανώθηκαν, 8.000 project ε, πήρανε την, το βραβείο της χρονιάς. Προσπαθήσαμε να φτάσουμε στην, στους νέους, γιατί πραγματικά αυτούς αφορά η πολιτική κληρονομιά. Ένα project είναι το Discovery U, μια πιλωτική προτεραιότητα που ξεκίνησε από την Κομισιόν Φέτο με, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 15.000 νέοι Ευρωπαίοι έλαβαν ελεύθερα, ε, ελεύθερο πάσο δωρεάν για να ε, ανακαλύψουν την πολιτική κληρονομιά της Ευρώπης, για να μάθουν από άλλους νέους και να ανταλλάξουν εμπειρίε για το τι σημαίνει να είναι κανεί Ευρωπαίος. Δύο από αυτούς ε, αποτέλεσαν τους ερευνητές της χρονιάς για την πολιτιστική κληρονομιά με post στα ε, μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το τι σημαίνει πολιτιστική κληρονομιά και καλώντας τους ε, φίλους τους να ε, ωφεληθούν από αυτή την ευκαιρία. Επίσης, πάλι για το Ευρωπαϊκό Έτος, ήταν οι διάφοροι χάρτες που εκπονήθηκαν από το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης online πλατφόρμα αυτή ε, που βάζει την, ε, ε, ουσιαστικά που φέρνει πιο κοντά την πολιτική κληρονομιά στους πολίτες με πολύ εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες για διάφορες πρωτοβουλίες τις οποίες διεξάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η εταίροι της προς όφελος της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς όπως το, το βραβείο της Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς. Επίσης, πρόσβαση στις ψηφιακές συλλογές της Europeana που περιλαμβάνουν πάνω από 50 εκατομμύρια έργα βιβλία από 3.500 πολιτιστικά ε, ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη. Μέχρι στιγμής οι χάρτες αυτοί έχουν ε, φτάσει σε 15.000 ε, χρήστες και καθημερινά προσπαθούμε το νούμερο αυτό να αυξηθεί. Αυτά τα νούμερα είναι πολύ ενθαρρυντικά και αποτελούν μια σύγκληση ανθρώπων από όλη την Ευρώπη που θέλουν να ανακαλύψουν εκ νέου την Ευρώπη και την πολιτιστική της κληρονομιά δραστηριότητες που έγιναν σε, από τις μικρότερες περιοχές μέχρι τις μεγαλύτερες πόλεις. Επαναλαμβάνουν την δέσμευση των πολιτών προς την ευρωπαϊκή κληρονομιά και την, το κοινού μας χώρου. Ένα παράδειγμα είναι οι, ε, οι καμπάνες που ήχησαν ε, για την Διεθνή ημέρα ειρήνης. 21 Σεπτεμβρίου ήχησαν καμπάνες σε εκκλησίες, σε δημαρχία, σε 14 ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η συμβολική πράξη μας θυμίζει ότι παρόλο που μιλούμε διαφορετικές γλώσσες, έχουμε διαφορετικές ιστορίες και διαφορετικές απόψεις, ο ήχος των, ε, των καμπανών ε, μεταδίδει ένα ε, παρανθρώπινο μήνυμα για το μέλλον. Εγώ βλέπω πώς αυτές οι εμπειρίες επιτρέπουν στους πολίτες να εξετάσουν και την τοπική τους ταυτότητα, την εθνική τους ταυτότητα μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Έτσι μόνο μπορούμε να αναγνωρίσουμε την, το, τις επικαλύψεις που υπάρχουν μέσω των ταυτοτήτων μας και των κοινωνιών μας. Πιστεύω και πιστεύω ότι το ξέρετε κι εσείς ότι έχουμε μια κοινή ιστορική εμπειρία και αναγνωρίζοντας αυτό μπορούμε πραγματικά να προχωρήσουμε δεδομένων και των εντάσεων που υπάρχουν τώρα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό θα ήταν λοιπόν να θυμόμαστε το πιο θεμελιώδης δίδαγμα από αυτή τη χρονιά. Υπάρχουν πολύ περισσότερα που μας ενώνουν από αυτά που μας χωρίζουν. Αυτή η αίσθηση ενότητα πραγματικά χαρακτηρίζει το ευρωπαϊκό Έτο. Είναι πολύ μεγάλη, μεγάλου φάσματος σε πρωτοβουλία, περιλαμβάνει όλα τα θεσμικά όργανα, όλα τα κρατημέλη της Ένωσης, εννέα χώρε εταίρους και επίσης ε, πάρα πολλούς εμπλεκόμενους εθνικούς φορείς. Είδαμε την στήριξη και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρηματοδοτεί με 800.000 ευρώ ένα πιλωτικό πρόγραμμα για την ε, ε, διερεύνηση ε, ε, των εβραϊκών νεκροταφείων σε πέντε χώρες. Επίσης καταγράφονται οι καλές πρακτικές για, την, ε, για τα εβραϊκά νεκροταφεία και προτείνεται και ένα μοντέλο για την διασφάλισή τους μέσω των τοπικών κοινοτήτων. Γιατί είναι σημαντικό αυτό στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έτους. Γιατί αυτά τα νεκροταφεία αποτελούν μία από τις, από τους, έναν από τους χώρους που απειλήθηκαν μεταξύ άλλων ιστορικών χώρων. Ε, εγγυόμενοι λοιπόν την ε, αποκατάστασή τους μπορούμε να καθοδηγήσουμε τους ε, νέους μας και να καθοδηγηθούμε και εμείς στην καθημερινή μας ζωή. Αυτό επίσης φαίνεται και στις προπαρασκευαστικές δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρόθεση καινοτόμων επιχειρησιακών μοντέλων για υγιή ε, σπίτια στην ε, ε, Ευρώπη. Το 40% των οικημάτων βρίσκεται σε ιδιωτικά χέρια. Για να μπορέσουμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε το μέλλον αυτών των κτηρίων θα πρέπει να δούμε πώς ήταν η ζωή για τους προγόνους μας και να δούμε πώς έχουμε προχωρήσει. Κυρίες και κύριοι. Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα ολοκληρωθεί σε λίγε εβδομάδε, αλλά εμεί θα φροντίσουμε η ευρωπαϊκή κληρονομιά να παραμείνει στο κέντρο τη Ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα. Το Μάιο έκανα μια πρόταση για μια νέα, ένα νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τον πολιτισμό με βασικό σημείο την αναγνώριση του πολιτισμού και της ποικιλομορφίας του πολιτισμού ώστε η Ευρώπη να γίνει κοινωνικά πιο συνεκτική και πιο ανταγωνιστική να μας βοηθήσει να έχουμε καλύτερους δεσμούς με τους εταίρους μα σε όλο τον κόσμο. Ένα βασικό πυλώνα του θεματολογίου είναι ένα σχέδιο δράση για την πολιτιστική κληρονομιά, το οποίο θα ε, ε, παρουσιάσω στι 7 Δεκεμβρίου στην επίσημη διάσκεψη για το κλείσιμο του Ευρωπαϊκού Έτου στη Βιέννη. Αυτό το σχέδιο δράση θα ορίσει μια ε, κληρονομιά πολιτικών για το Ευρωπαϊκό Έτο και θα αποτελέσει και έναν οδικό χάρτη για τη μελλοντική μα δουλειά για τη διασφάλιση και προώθηση τη πολιτιστική κληρονομιά τη Ευρώπη. Θα ξεκινήσει από δράσει όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει κατά τη διάρκεια του έτου, σύμφωνα και με τι αρχέ της ε, βιωσιμότητας, της προστασίας και της καινοτομίας. Θα καλύπτει θέματα όπως ε, η νεολαία, προσβασιμότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς και δραστηριότητες για να αντιμετωπίσουμε το παράνομο εμπόριο πολιτιστικών αγαθών. Καινοτομία και επιστήμες επίσης, πολύ σημαντικός ε, τομέας το σχέδιο δράσης θα αποτελέσει και την έμπνευση για τις περιφέρειες και τις πόλεις της Ευρώπης, αλλά και για τις οργανώσεις πολιτιστική κληρονομιάς και για τα σχετικά δίκτυα όταν εκπονούν τις δικέ τους δράσεις για την πολιτιστική κληρονομιά. Δεν μπορεί να υπάρχει πολιτική χωρί βεβαίω να υπάρξει απαραίτητη χρηματοδότηση. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί ο, πολιτισμό. Ε, ο προπολογισμό ε, του Creative Europe στο 1,85 δις ευρώ για την επόμενη περίοδο μέχρι το 2020. Οι διαπραγματεύσει για τον προπολογισμό εξελίσσονται και βεβαίω πάντα υπάρχουν προβλήματα και προκλήσει. Αυτή λοιπόν είναι μια στιγμή για όλου μα. Όσου πιστεύουν στον, ε, στη δύναμη τη πολιτική κληρονομιά, ότι μπορεί να δημιουργήσει μια πιο συμμετοχική Ευρώπη, ότι μπορούμε να σταθούμε όλοι δίπλα ο ένα τον άλλον και να την προωθήσουμε. Με τη στήριξή σα είμαι σίγουρο ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. Σα ευχαριστώ και πάλι για τη σκληρή δουλειά σας και βεβαίως προσβλέπω να σας δω όλους ή πολλούς από εσά στην ε, διάσκεψη στη Βιέννη. Σας ευχαριστώ. vielen herzlichen Dank. Εγώ ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα συμφωνήσω με αυτά που είπατε και θα χρησιμοποιήσω και την ευκαιρία αυτή για να σας ευχαριστήσω και εγώ όλους. Ευχαριστώ που συμμετείχατε τόσο ενεργά σε αυτή την ε, διήμερη διάσκεψη εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σας ευχαριστώ που με τις παρεμβάσεις σας δείξατε ότι το έτος ε, πολιτιστικής κληρονομιάς θα ε, δείξει τον αντίκτυπό του και μετά το έτος του 2018. Αυτό πιστεύω ότι είναι η μεγαλύτερη επιτυχία αυτής της πολιτιστικής πρωτοβουλίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν θέλουμε βεβαίως να διασφαλίσουμε μια βιωσιμότητα αυτού του project. Χωρίς λοιπόν τώρα άλλες καθυστερήσεις, κλείνουμε τη σημερινή διάσκεψη. Ευχαριστώ όλους τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων, τους συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ευχαριστώ όλους τους προσκεκλημένους φορείς και σας καλώ όλους σε ένα μικρό κοκτέιλ στην, στο εστιατόριο στον τρίτο όροφο. Οπότε εκεί θα μπορέσουμε να εμβαθύνουμε τις συζητήσεις μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν όλοι παρόντες σήμερα. Η Πρόεδρος ευχαριστεί και τους Δερμηνείς. Ευχαριστώ όλους και υπάρχουν και υπάρχει ενημερωτικό υλικό με φυλάδια, με μελέτες και τα λοιπά έξω από την αίθουσα και επίσης μια οικογενειακή φωτογραφία που πρέπει να βγάλουμε εδώ μπροστά στο Προεδρείο. Οπότε ελάτε όλοι εδώ για να βγάλουμε πρώτα τη φωτογραφία και μετά να πάμε στο κοκτέιλ. Ευχαριστώ όλους και για τα μέλη της Επιτροπής θα λέμε το απόγευμα.